so Αγαπητοί συνάδελφοι, αρχίζουμε τη συνεδρίασή μας παρά το γεγονός ότι είμαστε πολύ λίγοι, αλλά αυτοί που πραγματικά ενδιαφέρονται είναι παρόντες. Αρχίζουμε με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι μία ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Πίτερ Τόμσον, ο οποίος είναι πρόεδρος ε, των Ηνωμένων Εθνών, της ε, ε, Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και ασχολείται με την βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους της χιλιετίας. Και αυτό σε σχέση με τους στόχους της χιλιετίας και τους αναπτυξιακούς στόχους θα ήθελα να καλωσορίσω τον πρόεδρο Τόμσον που ήρθε στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε πολύ που ε, μεταβήκατε εδώ στις Βρυξέλλες και θα μας πείτε πώς έχουν ε, εξελιχθεί οι βιώσιμοι αναπτυξιακοί στόχοι, γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλουμε προσπάθειες επί του θέματος. Επίσης, ε, μας ενδιαφέρει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η διάσκεψη των ωκεανών που θα διεξαχθεί τον Ιούνιο. Και σας δίνω το λόγο άμεσα. Thank you very much, um, and uh, Mr. Chairman and uh, uh distinguished members Ευχαριστώ πολύ αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου. Ε, σας ευχαριστώ για όλα τα καλά σας λόγια και είναι μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι σήμερα εδώ στην Επιτροπή. Θα ήθελα να ευχαριστώ την Επιτροπή που μου δίνει τη δυνατότητα να συναντηθώ με τα μέλη της Επιτροπής ε, και ε, φαντάζομαι ότι στις σημερινές συνεδρίες μπορούν να συμμετέχουν και βουλευτές από άλλε επιτροπές. Κυρίε και κύριοι, κάθε μέρα η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις. Ε, προκλήσεις που είναι πολύ περίπλοκες. Ε, ξεκινάνε από θέματα που έχουν σχέση με την διεθνή ειρήνη και την ασφάλεια και φτάνουν μέχρι στη μεγαλύτερη μεταναστευτική κρίση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βλέπουμε την εξάπλωση τη τρομοκρατίας και βίες ακραίες πράξεις έναντι 125 ε, εκατομμυρίων ανθρώπων. Εμείς επιθυμούμε να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των δύο φύλων και προσπαθούμε βεβαίως και να προστατεύσουμε το κλίμα σε ολόκληρο τον κόσμο. Αναμφίβολα όλα αυτά τα θέματα που συζητούνται σήμερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλονται κυρίως στο ότι υπάρχουν ε, πρωτοφανείς ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο η Ευρώπη και ο πλανήτης μας. Η Ευρώπη πλήττεται από την τρομοκρατία, από τις ροές των μεταναστών, των προσφύγων, αλλά υπάρχουν και πολιτικές αναταραχές που προκύπτουν από μια εποχή μεγάλης ανασφάλειας. Το να αντιμετωπίσει κανείς αυτές τις παγκόσμιες προκλήσεις, αυτό προϋποθέτει την ενότητα και την αλληλεγγύη, γιατί οι κοινέ προκλήσεις απαιτούν και συλλογικέ απαντήσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την ευγνωμοσύνη μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το ότι έχει συμβάλει στην ε, διεθνή ανάπτυξη γιατί είναι ένας μεγάλος ανθρωπιστικός παίκτη. Το πνεύμα αυτό ε, θα πρέπει να συνεχίσει να επικρατεί στις προσπάθειές μας. Όλοι μας, μονομενά άτομα, κοινότητες, ε, κράτη, όλοι μας καλούμεθα να αναζητήσουμε παγκόσμιες λύσεις έτσι ώστε να επιτύχουμε το μέλλον μας που θα είναι ασφαλές και με ευημερία για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Κυρίες και κύριοι, η ατζέντα της βιώσιμης ανάπτυξης του 2030 μας δίδει ε, ένα πρόγραμμα για το μέλλον, η αποτελεσματική εφαρμογή της ε, ατζέντα του 2030 από κοινού με τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Αυτά θα αλλάξουν τον κόσμο, θα εξαλείψουν την ακραία φτώχεια και θα προωθήσουν την ισότητα των δύο φύλων, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου και του ωκεανού. Θα αποτελεσματικά η κλιματική αλλαγή. Η ατζέντα και οι 17 στόχοι της ε, χιλιετίας είναι φιλόδοξοι και πρέπει να είναι. Εξετάζοντας λοιπόν αυτές τις ε, δεσμεύσεις μας, αυτό απαιτεί από όλους τους εταίρους, από τις κυβερνήσεις, τα Ενωμένα Έθνη, περιφερειακούς και πολυμερείς οργανισμούς, από την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα, από την επιστημονική και την φιλανθρωπική κοινότητα, όλοι να συνεργαστούν για να εφαρμοστούν οι στόχοι της χιλιετίας. Και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο, πρώτον προάγοντας τον οικουμενικό χαρακτήρα των στόχων της χιλιετίας, και διασφαλίζοντα ότι αυτοί βρίσκονται μέσα στα όρια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση, χρησιμοποιώντα τα διάφορα εργαλεία που έχει και τι πολιτικέ, τι προδιαγραφέ τη αγοράς, ε, την υποδομή, τι ενεργειακέ πολιτικέ, μπορεί να στηρίξει την εφαρμογή των στόχων τη Χιλίτια. Και τρίτον, αν ε, μπορέσουμε να επιτύχουμε το 0,7 του ΑΕΠ για τι δεσμεύσει μα, θα μπορέσουμε με τον τρόπο αυτό να προσφέρουμε υποστήριξη στου ε, στόχου τη χιλιετίας σε όλες τις χώρες του κόσμου. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ότι επιδεικνύει καθοδηγητικό πνεύμα στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη έχουν καταβάλει προσπάθειες για να προάγουν την εφαρμογή των στόχων της χιλιετίας και τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Και εδώ περιλαμβάνεται και η εργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να υπενθυμίζει σε όλους τους θεσμούς και στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις υποχρεώσεις τους ε, και τις ενέργειες που οφείλουν να αναλάβουν. Κυρίε και κύριοι, εάν κατορθώσουμε να προχωρήσουμε με ταχύτητα και να επιτύχουμε τους στόχους της χιλιετίας μέχρι το 2030, για να γίνει αυτό πρέπει να λάβουν χώρα και ορισμένα βασικά βήματα. Ορισμένα εξ αυτών έχουν μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να υπάρξουν καινούριε, καινοτόμε στρατηγικές συνεργασίες και επίσης να χρησιμοποιήσουμε την καινοτομία και την τεχνολογία που είναι καταλητικοί παράγοντες για να επιτύχουμε βιώσιμη ειρήνη και ανάπτυξη. Οφείλουμε από τη γραμμική πρόοδο στην τεχνολογία να περάσουμε σε εκθετική πρόοδο. Ενώ λοιπόν έχουμε κατά νου την τεχνολογία και τις μεθόδους που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργηθούν θέσεις απασχόληση, θα ήθελα να καλέσω όλους σας να εξετάσετε το πώς μπορεί κανείς να δαμάσει τις νέες τεχνολογίες για να προσφέρει περισσότερες ε, περισσότερη υποστήριξη στη βιώσιμη παραγωγή. Ε, ο πληθυσμός του κόσμου αυξάνεται και γι' αυτό οφείλουμε να κινητοποιήσουμε όλες μας δυνάμεις αν θέλουμε να επιτύχουμε τους στόχους της χιλιετίας. Αυτό λοιπόν προϋποθέτει την μεταρρύθμιση της παγκόσμιας οικονομίας. Πριν από δύο ημέρες είχαμε σχετικές συζητήσεις επί του θέματος και εγώ συνεκάλασα ε, στα κεντρικά γραφεία των ΗΕ μία συνάντηση υψηλού επίπεδου. Μεταξύ άλλων καταλήξαμε στο ότι είναι απαραίτητο να χρηματοδοτήσουμε τους ε, ήδη βιστάμενους στόχους της χιλιετίας σε ολόκληρο τον κόσμο και αυτά να προσαρμοστούν με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Δεύτερον, ενώ οι στόχοι της χιλιετίας έχουν νόημα οικονομικά για τις επιχειρήσεις, με την εφαρμογή των στόχων της χιλιετίας μπορούν να προκύψουν εκατομμύρια δολαρίων που θα τοποθετηθούν στην αγορά και βέβαια παράλληλα μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερα για να συνδυάσουμε την χρηματοδότηση με βιώσιμα και από τις τράπεζες επιλέξιμα προγράμματα. Κυρίες και κύριοι, Νομίζω ότι ε, θα ήθελα να σας ενταρρύνω όλοι μας να επιδιώξουμε τους στόχους της, ε, του θεματολογίου 2030. Το θεματολόγιο αυτό θα μπορεί να έχει πολύ σημαντικές ε, επιπτώσεις. Όσον αφορά εμένα, εγώ θα ήθελα να ε, φέρω κοντά τους παίκτες, ε, να διαδώσω τις κοινέ μας απόψεις και να ενισχύσω τις προσπάθειες για να εφαρμοστούν και οι 17 στόχοι της χιλίτιας. Και προς αυτή την κατεύθυνση έχω καλέσει μια σειρά, συγκαλέσει μια σειρά ε, συνεδριάσεων υψηλού επίπεδου με θέμα, όπως σας είπα, την στήριξη της ειρήνης, την κλιματική αλλαγή και τα θέματα τα χρηματοπιστωτικά. Η επόμενη συνάντηση θα λάβει χώρα στις 17 Μαΐου και θα έχει ως θέμα την καινοτομία και την ε, διασύνδεση, την connectivity. Υπάρχουν όμως κυρίες και κύριοι και άλλα δύο θέματα τα οποία θα ήθελα να σας επισημάνω. Αυτά θα είναι μεγάλη σημασία στη Γενική Συνέλευση των ΗΕ που θα λάβει η χώρα κατά τους επόμενους μήνες. Το πρώτο έχει σχέση με την ε, συνδιάσκεψη για τους ωκεανούς θα λάβει χώρα μετά από ένα μήνα. Ε, θα συναντηθούν πολλοί εκπρόσωποι από ολόκληρο τον κόσμο στη Νέα Υόρκη. Αναφέρομαι κυρίως εκπροσώπους της ε, ανθρωπότητας, γιατί θα έχουμε βεβαίως αρχηγούς κρατών, ε, κυβερνήσεων, υπουργούς ε, που θα παρίστανται, αλλά θα συμμετέχουν και πυρογνώμονες για τον ωκεανό, ακτιβιστές και παΐοντες από τον ιδιωτικό τομέα, την κοινωνία των πολιτών, τις ΜΚΟ, τον ακαδημαϊκό χώρο και την επιστημονική κοινότητα. Για πέντε ολόκληρε ημέρες, από τις 5 μέχρι τι 9 Ιουνίου, θα έχουμε 150 παράλληλες συνεδριάσεις, επίσης 7 ε, διαλόγους που θα έχουν συγκεκριμένο στόχο που θα είναι οι στόχοι της χιλιετίας, ο συγκεκριμένο υπαριθμό 14 που αφορά τους ωκεανούς. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας πω ότι οι ωκεανοί αντιμετωπίζουν προβλήματα. Γνωρίζετε όλοι ότι υπάρχουν καταστροφικές αλλιευτικές πρακτικές, καταραίουν τα αλλιευτικά αποθέματα και σε κάποια στιγμή φοβάμαι μέχρι το 2050 θα έχουμε περισσότερα πλαστικά προϊόντα στους ωκεανούς παρά ψάρια. Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε σχέση με τους ωκεανούς. Ο κατάλογος είναι μακροσκελής και όπως σας είπα θα συγκληθεί η συνάντηση αυτή ως το μόνο παγκόσμιο φόρουμ το οποίο θα έχει ως στόχο να κινητοποιήσει τον κόσμο για να αντιμετωπίσει την ε, ε, τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουν προκύψει κυρίως σε σχέση με το στόχο υπερθμών 14 των στόχων της χιλιετίας. Πέρα λοιπόν από την παγκόσμια ευαισθητοποίηση για την καταστροφική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Ακεανοί, θα έχουμε και άλλους τρεις στόχους. Πρώτον, ε, έκκληση για πρόγραμμα δράσης ε, η διατύπωση αυτού του προγράμματος δράσης θα είναι απόλυτα ακριβής. Κατά δεύτερον θα υπάρξει μια έκθεση πάλι για δράσεις και λύσεις ε, που θα προκύπτουν από τους 7 διαλόγους που θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο της ε, συνδιάσκεψης. Κάθε ένας εξ αυτών θα αφορά ένα συγκεκριμένο στόχο της χιλιτίας που θα έχει σχέση με τη ρήπανση, με τη διαχείριση των ωκεανών. Τρίτον, ε, θα υπάρξει καταγραφή των ε, προαιρετικών δεσμεύσεων, δηλαδή θα καταγραφούν όλοι εκείνοι που δεσμεύονται να στηρίξουν το στόχο των υπαριθμών 14 και να συμβάλλουν στη διαφύλαξη της ζωής του ωκεανούς. Η ε, εθελοντική δέσμευση αυτή μπορεί να υπάρξει μέσα από την ιστοσελίδα της ε, συνδιάσκεψη. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, την ώρα, μέχρι την ώρα που θα λάβει η χώρα η συνδιάσκεψη να έχουμε πολλούς ατελεντοές γιατί έτσι θα εκπροσωπούνται και όλες οι εκφάνσεις ε, που έχουν σχέση με το στόχο υπαριθμών 14. Είμαι σίγουρος ότι τα κράτη-μέλη θα συμμετάσχουν στη συνδιάσκεψη, καλό και εσά τους βουλευτές να είσαστε παρόντες. Επίσης θα ήθελα και στις εκλογικές περιφέρειες, να απευθυνθείτε σε τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνία των πολιτών, σε επιχειρήσεις, να καταγραφούν και αυτοί στους εθελοντές στην ιστοσελίδα της συνδιάσκεψης για τους ωκεανούς. Τώρα είναι κατάλληλη στιγμή για καταγραφή, για να ξέρουμε ποιοι θα δραστηριοποιηθούν για να επιτύχουμε τον ευγενή στόχο υπαρτμών 14. Κυρίες και κύριοι, το δεύτερο θέμα το οποίο θέλω να σας επισημάνω είναι η μετανάστευση. Για να επιτευχθούν οι στόχοι της χιλιετίας τα επόμενα 14 χρόνια, πρέπει να προβούμε και σε χρηματοδότηση επιτόπου. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι τα ωφέλη της βιώσιμη ανάπτυξης θα φτάσουν σε όλους, δεν θα εξαιρεθεί κανείς. Το όλοι σημαίνει κυρίως τα περιτυροποιημένα και ευάλωτα μέλωτα, μέλη της κοινωνίας μας, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των μεταναστών. Σε ολόκληρο τον κόσμο ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί πρόσφυγες και μετανάστες οι οποίοι υφίστανται το ρατσισμό, την ξενοφοβία, την μυσαλλοδοξία. Ε, απομονώνονται ε, αποκλείονται από εκπαιδευτικές ευκαιρίες και καλούνται να ζήσουν την διάκριση στο πετσί τους. Για να αντιμετωπιστούν λοιπόν όλες αυτές οι προκλήσεις, τα κράτη-μέλη των ΗΕ εργάζονται και προσπαθούν να βελτιώσουν την παγκόσμια διαχείριση, να ενισχύσουν τη διεθνή συνεργασία για θέματα μετανάστευσης. Η προετοιμασία έτσι ώστε να έχουμε ασφαλείς ροές μεταναστών, όπως επίσης και θετικές, θετικό αντίκτυπο στους πρόσφυγες, όλα αυτά έχουν ήδη ξεκινήσει και προσβλέπουμε σε πάρα πολλά. Ενδεχομένως θα γνωρίζετε ότι κατά τους επόμενους έξι μήνες θα οργανώσουμε μία σειρά θεματικών συζητήσεων με ε, παγκόσμιο αντίκτυπο. Αυτά θα λάβουν χώρα στη Νέα Υόρκη, τη Γενέβη και τη Βιέννη. Και θα ακολουθήσει μία προκατακτική συνάντηση το Δεκέμβρη στο Μεξικό. Μετά από αυτή τη συνάντηση θα παρουσιαστεί ένα σχέδιο για τη μετανάστευση. Αυτό θα συμβεί το 2018 και θα παρουσιαστεί το σχέδιο στα κράτη-μέλη για να εγκριθεί σε μια δικυβερνητική συνδιάσκεψη που ελπίζουμε να λάβει η χώρα πριν από τη γενική συζήτηση σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών. Κυρίες και κύριοι, εσείς ε, ως ε, ξέχουσες προσωπικότητες και ευρωβουλευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε ισχυρή φωνή. Σας καλώ λοιπόν να χρησιμοποιείτε τις ε, πλατφόρμες μας, να μας στηρίζετε σε όλα αυτά τα δύσκολα και κρίσιμα θέματα που πιο κρίσιμο δεν υπάρχει από, την, ε, ε, το θεματολόγιο του 2030 για την βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτή είναι η ελπίδα μας για να διασφαλίσουμε την ανθρωπιά στον κόσμο. Ο Ότο Φον Μπίσμαρκ, μεγάλος ηγέτης του 19ου αιώνα, μα είπε ότι η διαφορά ανάμεσα ένα πολιτικό και έναν κυβερνώντα είναι ότι οι πολιτικοί έχουν κατά νου κυρίως την ευημερία των απογόνων τους. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ θα ήθελα να συμβάλλετε κι εσείς έτσι ώστε να επιτύχουμε την αποτελεσματική εφαρμογή του θεματολογίου του 2030 τόσο στην Ευρώπη όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Your Excellency, ε, σας ευχαριστώ για τα πολύ σημαντικά λόγια σας ε, που μας εμπνέουν και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας υποστηρίξουμε. Τώρα θέλω να καλέσω τους συναδέλφους που θέλουν να συμμετάσχουν στην συζήτηση να πάρουν το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, λέει ο Ζαβόρ. Ε, ευχαριστώ, κύριε Τόμσον, για την παρουσίασή σας. Θα ήθελα να μιλήσω λιγάκι για την εφαρμογή των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είμαι υπεύθυνο για τη σχετική νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να αναφέρω πέντε βασικά σημεία που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη σωστή εφαρμογή των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρώτο που εγώ πιστεύω ότι πρέπει να εφαρμοστεί σωστά ο πρώτος από τους 17 στόχους ε, και τους 169 επιμέρους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης είναι η ανάγκη για μια συνολική ε, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή των στόχων. Ε, αν μιλήσουμε για το ένα ε, αποκομμένα από τα υπόλοιπα, δεν νομίζω ότι θα καταφέρουμε ας πούμε, να πετύχουμε τους περιβαλλοντικούς στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης χώρια από τους άλλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει περισσότερα και να δεχθεί ε, μια συνολική στρατηγική για να προωθήσει συνολικά τους στόχους ε, και να ελέγχει τις ισχύουσες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τους αντιπαραβάλλει με τους ε, στόχους τη βιώσιμης ανάπτυξης και να βλέπει αν οι πολιτικές συνεισφέρουν στην εφαρμογή των στόχων ή αν είναι κατά και μας εμποδίζουν να του υλοποιήσουμε αυτού τους στόχους. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη τις κοινωνικέ πτυχέ. όπως πρέπει, σωστά. Κυρίω να δώσουμε προσοχή στι ευάλωτε ομάδε πληθυσμού. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικέ φορές έχω την αίσθηση ότι αυτοί οι στόχοι έχουν ένα περιβαλλοντικό, μια περιβαλλοντική πτυχή που είναι σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα για την ε, βιωσιμότητα και το περιβαλλοντικό κομμάτι της βιωσιμότητας, αλλά το κοινωνικό τμήμα, ε, η πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες, θεωρούμε ότι αυτό είναι θέμα των χωρών του Νότου, τρίτων χωρών, άλλων. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν εκατομμύρια εκατομμυρίων Ευρωπαίοι που ζουν σε βαθιά ένδια, ε, που δεν έχουν πρόσβαση στο νερό, που δεν έχουν ε, πρόσβαση στην αποχέτευση, δεν έχουν σωστή ε, περίθαλψη, δεν έχουν σωστή στέγη, ενέργεια κλπ. κλπ. Επομένως και κοινωνικά πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κοινωνικοί στόχοι των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και οι επιμέρους κοινωνικοί στόχοι πρέπει να υλοποιηθούν, γιατί εκατομμύρια Ευρωπαίων δεν έχουν αυτό που θα έπρεπε να έχουν. Το τρίτο βασικό στοιχείο, και το αναφέρατε και εσείς κύριε Τόμψον, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η επαρκής χρηματοδότηση. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο θα δοθούν πραγματικά οι κατάλληλοι πόροι για την εφαρμογή αυτών των στόχων, αλλά συστηματικά θα πρέπει να ελέγχουμε όλο το, όλα τα δημόσια κονδύλια και αν συνάδουν με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Γιατί μερικές φορές παταλάμε χρήματα ε, επιδοτώντας δραστηριότητες που δημιουργούν προβλήματα ε, και μετά με άλλες επιδοτήσεις πάλι από, τα δημόσια, από το δημόσιο κορβανά προσπαθούμε να καθαρίσουμε τις ε, συνέπειες της λάθος αρχικής χρηματοδότησης. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν συνεπείς στη χρηματοδότηση και θα πρέπει συστηματικά, να ελέγχουμε την ε, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και να αντιπαραβάλλουμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Και να μην ε, ε, δημιουργούμε υποδομές που κλειδώνουν τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά μας συστήματα σε μια πορεία μη βιωσιμότητας. Επίσης, το τρίτο και βασικό στοιχείο είναι η συμμετοχή των πολιτών και των ε, φορέων, η καλή διακυβέρνηση κατά την εφαρμογή των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Δεν νομίζω ότι είναι αρκετό το να δεχτούμε, το να έχουμε μια καλή νομοθεσία και να την εφαρμόσουμε. Δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να συμπεριλάβουμε και την κοινωνία. Η κοινωνία πρέπει να είναι τμήμα Τη ε, νομοθετικής διαδικασίας του σχεδιασμού και να είναι τμήμα προφανώς τη εφαρμογή. Γιατί αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε καλή διακυβέρνηση και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πείσουμε την κοινωνία ότι οι στόχοι της βιώσιμη ανάπτυξης είναι κάτι που τους αφορά, ε, που την αφορά, που αφορά του πολίτε. Και το τελευταίο βασικό σημείο, το πέμπτο, είναι η ανάγκη να μειώσουμε τι αρνητικέ επιπτώσει της κατανάλωσής μας, του τρόπου κατανάλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσφατα υιοθετήσαμε μία έκθεση δύο πρωτοβουλίας για το φινικέλαιο, που είναι ένα παράδειγμα τέτοιας κατανάλωσης. Ε, ότι μερικές φορές αυτά που καταναλώνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δημιουργούμε προβλήματα βιωσιμότητα μεν, δημιουργούμε όμω τεράστια προβλήματα βιωσιμότητα εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ο τρόπο κατανάλωση, η οικονομική και η κοινωνική λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο τι δικέ μα κοινωνίε, έχει τεράστιε επιπτώσει όμω και εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν θέλουμε πραγματικά να υλοποιήσουμε του στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη, θα πρέπει μονίμω να ελέγχουμε ε, αν επηρεάζουμε ε, εμείς με τον τρόπο που ζούμε και καταναλώνουμε ε, την εφαρμογή των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να τους προωθούμε και όχι να τους καταστρέφουμε. Κυρία Ντελάε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις στα πλαίσια της ε, διάσκεψης για τους ωκεανούς που θα γίνει σε λίγες εβδομάδες στη Νέα Υόρκη. Η πρώτη ερώτηση αφορά την, ε, τις θαλάσσιες ενέργειες ο ΙΕ στα πλαίσια της εφαρμογής των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, πώς προτίθεται να προωθήσει την ε, διατήρηση των πόρων κρατώντας τις θέσεις απασχόλησης. Γιατί φυσικά και αυτό είναι τμήμα των στόχων που πρέπει να σεβαστούμε. Δεύτερον, το δεύτερο αφορά τις ευρωπαϊκές περιφέρειες ε, που είναι νησιωτικές. Διερωτώ με, εάν προβλέπονται ειδικά μέτρα από τον ΟΗΕ για αυτές τις ε, περιοχές, για αυτές τις περιφέρειες, ούτω ώστε οι υπερπόντιες ε, περιοχές να ενταχθούν στα πλαίσια αυτά της ε, υλοποίησης των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Δύο απλές ερωτήσεις, πολύ άμεσες. Θα ήθελα να μου δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριος Φρόντε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για αυτή τη συνάντηση, που για μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Ειδικά για τους ωκεανούς. Εγώ, θα είμαι, εγώ είμαι τμήμα της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Περιβάλλοντος που θα πάει στην Νέα Υόρκη τον Ιούνιο. Και επίσης διοργανώνω και μια παράλληλη εκδήλωση που αφορά το Μάρι Λίτερ, το οποίο συζητάμε και εδώ στην Ευρώπη δηλαδή τη διαπραγμάτευση για τις θάλασσες. Αυτό συνδέεται με το στόχο 14, που αφορά και τους ωκεανούς. Καταρχάς, εμείς μιλάμε πάρα πολύ για την μπλε ανάπτυξη και για την μπλε οικονομία. Φυσικά, έχουμε τις καλύτερες προθέσεις όταν το συζητάμε για αυτά. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μία έρευνα από το ερευνητικό κέντρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Αλία και που μας έδειξε πώς από τη μία η μπλε ανάπτυξη θα δημιουργήσει περισσότερες θέσεις απασχόλησης και μεγαλύτερο ΑΕΠ, αλλά δημιουργεί πολλά ερωτηματικά σε ό,τι αφορά τις αρτικές συνέπειες στο περιβάλλον. Ε, που αυτή η υπερβολική μπλε ανάπτυξη μπορεί να έχει. Από την άλλη, πρέπει να δούμε πώς οι ωκεανοί ε, είναι ένας νέος πόρος, ένα νέο σύνορο οικονομικής φύσεως από τη μία, αλλά και φυσικών πόρων από την άλλη. Αλλά αν το αντιμετωπίσουμε όπως αντιμετωπίσαμε όλους τους πόρους μας, τους φυσικούς πόρους σε παγκόσμιο επίπεδο, οι παγκόσμιες ε, περιβαλλοντικές συνέπειες θα είναι δύσκολο να τις διαχειριστούμε. Και πολύ σωστά εκφράζεται αυτό στο στόχο 14, η ανησυχία δηλαδή για την κατάσταση των, των ωκεανών. Με αυτά τα δεδομένα είναι πάρα πολύ σημαντικό στο τέλος της διάσκεψης της Νέας Υόρκης να γίνει μια τελική διακήρυξη με μια πολύ ισχυρή δέσμευση για τους ωκεανούς. Σας ρωτάω λοιπόν, εάν έχετε κάποια ιδέα κυρίως για δύο σημεία που αφορούν το σημείο 14, το 14-2 και το 14-4. Το 14-2 είναι πολύ σημαντικό γιατί λέει να ενισχύσουμε την αντίσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και να λάβουμε δράσεις για να αποκαταστήσουμε τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Είναι, ένας ε, ε, είναι εύκολο να το γράψουμε αυτό, αλλά είναι πολύ δύσκολο να το, φάρουμε, να το βάλουμε σε εφαρμογή. Ε, γιατί θα πρέπει να έχουμε δράσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Και μην ξεχνάτε ότι η κατάσταση της, των ωκεανών, ειδικά στις παράκτιες περιοχές, γίνεται όλο και χειρότερη με ταχύτατους ρυθμούς. Το άλλο θέμα είναι η υπεραλίευση. Εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, δουλεύουμε στα πλαίσια της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Δεν είναι πολύ εύκολο αυτό. Ε, θα πρέπει μέχρι το 2020 να δούμε τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Είμαστε πολύ μακριά, δυστυχώ, ε, παρότι γίνονται σημαντικά βήματα. Διερωτώ αν αυτή η τεράστια προσπάθεια που κάνει η Ευρώπη ε, ακολουθείται σε παγκόσμιο επίπεδο από αντίστοιχα μέτρα ε, από άλλες περιοχές του κόσμου για να αντιμετωπιστεί αυτή η υπεραλίευση. Το ένα βασικό πρόβλημα, και όχι το μοναδικό φυσικό, είναι ε, αυτό το πρόβλημα ε, της υπεραλίευσης και οι ωκεανοί μας επιδεινώνονται λόγω αυτής. Δεν είναι φυσικά το μόνο πρόβλημα, δυστυχώ. δυστυχώς. Ευχαριστώ. herzliches guten Morgen auch von meiner Seite. Ähm, Καλημέρα σας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κυρίως η Επιτροπή μας. Ε, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που είμαστε διαφανείς και που ε, συζητήσεις και συναντήσεις όπως η σημερινή μεταδίδονται μέσω διαδικτύου. Από την άλλη όμως αυτό έχει και το μειονέκτημα ότι όσοι Ευρωπαίοι ενδιαφέρονται για τέτοιου είδους ε, θέματα μπορούμε βέβαια να παρακολουθήσουμε τη συζήτηση αλλά υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που αντί να έρθουν εδώ να λάβουν το λόγο, κάτω στα γραφεία τους ε, και παρακολουθούν από εκεί τη συζήτηση. Σας τα λέω αυτά για να ε, καταλήξω. Μην νομίζετε ότι σας παρακολουθούν μόνο αυτοί που βρίσκονται στην αίθουσα. Είναι και άλλοι στα γραφεία τους που σας ακούνε πολύ προσεκτικά. Ε, να πω λοιπόν το εξής, ότι υπάρχουν πολύ συχνά πολιτικοί οι οποίοι δηλώνουν ότι γνωρίζουν και είναι προσιλωμένοι στους στόχους της ε, χιλιετίας. Και ε, οι απόψεις τους όμως δυστυχώς πολλές φορές αποκλίνουν από αυτά που θεωρούμε εμείς ως στόχοι. Ε, εγώ αυτούς τους στόχους τους θεωρώ και ως μια έκκληση για δράση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία δεν επιδιώκουν τους στόχους της χιλίτιας. Εμείς είμαστε αναγκασμένοι ε, να απευθυνθούμε στα κράτη αυτά για να τα επαναφέρουμε στο σωστό δρόμο. Και θέλω να ρωτήσω, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών υπάρχει ένα είδος ελέγχου, υπάρχει ένα είδος διαδικασίας monitoring, όπου κράτη-μέλη ναι μεν ρηματικά δηλώνουν ότι είναι προσιλωμένα στους στόχους χιλίτιας, στην πράξη όμως πράττουν ακριβώς το αντίθετο. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα να επισημάνουμε ότι αυτά τα οποία συζητούνται σε τελική ανάλυση θα πρέπει να είναι σε απόλυτη συμφωνία με αυτά τα οποία έχει δηλώσει κανείς ότι περασπίζεται. Η κυρία Μάισνερ. Και εγώ ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επίσης ευχαριστώ πολύ για την ομιλία σας κύριε Τόμψεν. Λυπάμαι που καθυστέρησα γιατί έπρεπε να ψηφίσω σε μια άλλη επιτροπή. Ε, ξέρετε, το θέμα που θίξατε με ενδιαφέρει πάρα πολύ, όχι μόνο γιατί έχω ασχοληθεί με την ολοκληρωμένη πολιτική των θαλασσών και την πλέον ανάπτυξη, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και διότι στο Κοινοβούλιο έχουμε μια διακομματική επιτροπή η οποία επιλαμβάνεται γενικότερα της μπλε ανάπτυξης και αυτή η Επιτροπή ε, ενδιαφέρεται τόσο για την εξυγίανση θα πω των θαλασσών που είναι απαραίτητη όσο και για την υποστήριξη της έρευνας για να γίνεται καλύτερη χρήση των θαλασσών και των ωκεανών. Είμαι πεπισμένη ότι οι συνάδελφοι από την ομάδα μου ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το ότι επειδή ε, έχουμε όλο και αυξανόμενο πληθυσμό στον κόσμο, θα αποκτήσουν και οι οικειοανοί μεγαλύτερη σημασία. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι πρέπει από κοινού να προχωρήσουμε. Γνωρίζετε την ε, Ocean Governance Strategy, τη σχετική ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανακοίνωση για τους ωκεανούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό βήμα και βεβαίως οι Ευρωπαίοι ενδιαφέρονται να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων σε παγκόσμιο επίπεδο για να γίνουν περισσότερα στοιχεία γνωστά για τους ε, ωκεανούς. Ε, βεβαίως, όλους μας μας ε, ενδιαφέρει να συζητήσουμε το κατά πόσον θα είναι δυνατόν να υπάρχει εξόριξη ορυκτών από το βυθό της θάλασσας. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει αυτό, θα καταστεί δυνατόν και είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη διαδικασία της εξόριξης να μην καταστραφεί η βιοπικιλότητα. Γιατί, ξέρετε, στη θάλασσα μπορεί να προκύψει πολύ μεγαλύτερη ζημιά από σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Στις θάλασσες και στους ωκεανούς δεν έχουμε μόνο πλαστικά προϊόντα, έχουμε την υπεροξίνηση, έχουμε ασθένειες ε, οι οποίε ε, ξεκινούν από τη θάλασσα και δεν ξέρουμε καθόλου το τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Εξάλλου και ολόκληρα νησιά ε, χάνονται, εξαφανίζονται λόγω της αύξησης της στάθμης της θάλασσα. Ε, πολλοί τα γνωρίζουν αυτά. Έχω πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις να σας κάνω. Δυστυχώς δεν άφησα την ομιλία σας. Θα ήθελα να σας ερωτήσω συγκεκριμένο σχετικά με τη διαχείριση των ωκεανών που υπάρχει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωση, Γιατί εκεί προτείνεται να υπάρχει κάποια παγκόσμια τάξη πραγμάτων που να αφορά όλους τους ωκεανούς. Εσείς τι πιστεύετε γι' αυτό. Ε, γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει κάποια ε, διάταξη, υπάρχουν κανόνες ε, για τη χρήση των θαλασσών και για το τι θα γίνει στο μέλλον. Αυτά λοιπόν που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις θάλασσες πιστεύετε ότι μπορούν να επεκταθούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Και επίσης ε, πιστεύετε ότι οι κανόνες θα μπορούσαν να υπογραφούν και από περισσότερες χώρες, γιατί αρκετές χώρες έχουν υπογράψει, αλλά δεν εφαρμόζουν τους κανόνες στην πράξη. Και νομίζω ότι αυτό είναι μία παράληψη για την υγιή εξέλιξη των ωκεανών. Και τρίτη ερώτησή μου, ξέρετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζουμε περισσότερο τις ε, έρευνες ε, στους ωκεανούς. Ε, δηλαδή όσοι ενδιαφέρονται αυτά γνωρίζουν ότι μιλάμε για μικτούς ωκεανούς και υπάρχουν συγκεκριμένα καθήκοντα που αφορούν στο μέλλον. Εσείς έχετε έτσι μια συγκεκριμένη εικόνα σχετικά με την έρευνα. Τι μπορεί να ενισχυθεί στην έρευνα πάντα σε σχέση με τις θάλασσες και τους ωκεανούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τώρα θα θα ήθελα ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να λάβει το λόγο, ο κύριος Ρίσε. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και εσάς, Πρόεδρε, της ε, Γενικής Συνέλευσης για την παρουσίασή σας. Η διάσκεψη των ωκεανών των Ηνωμένων Εθνών που θα λάβει η χώρα τον Ιούνιο είναι ένα μείζον γεγονός που δείχνει τη σημασία που προσδίδει η διεθνής κοινότητα στους ωκεανούς για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπέρ της Ατζέντα 2030 και θέλουμε να επιτύχουμε τον στόχο υπαριθμών 14, καθώς και όλους τους άλλους στόχους που σχετίζονται με τους ωκεανούς. Επίσης θέλουμε να ενισχύσουμε την διακυβέρνηση των ωκεανών. Έχει ήδη υποθεί ότι χρειάζεται μία στρατηγική υπέρ των νέων με κατευθυντηρίες γραμμές ως προς τις μελλοντικές πολιτικές σε αυτό το τομέα. Αυτή η διάσκεψη θα έχει μεγάλη σημασία για να προωθήσουμε τις συνεκτικές μας πολιτικές. Ο Επίτροπος Βέλα θα συμμετάσχει σε αυτή τη διάσκεψη. Την προπαρασκευάζουμε τώρα και έχουμε παρευρεθεί σε συναντήσεις ε, μέσα στα πλαίσια της έκκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος και δράσης για την ε, συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον διάλογο αυτό. Επίσης, τον Οκτώβριο ζητήσαμε μια άλλη διάσκεψη για τους ωκεανούς και υπάρχει συμπληρωματικότητα των δύο αυτών διασκέψεων. Γιατί ο ωκεανός και οι ωκεανοί είναι αναπόσπαστο μέρος της ανθρωπότητας. Κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε σε αυτό το λεπτό θέμα της μετανάστευσης. Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά τελευταία χρόνια, ειδικά πέρσι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης. Βεβαίως αυτό δεν είναι δυνατόν χωρίς τη δική σας συνεργασία και προσμένουμε στην πρόοδο και συνεργασία από τη δική σας πλευρά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη μετανάστευση και σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών σε σχέση με τον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης υπαριθμών 14 θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την κοινωνική διάσταση, την ε, συνολική μας στρατηγική και την επαρκή χρηματοδότηση για να υπάρξει μια επιπρόσθετη χρηματοδότηση και συνοχή καθώς και ένας ορίζοντας για τα συναφή αυτά θέματα. Ξέρετε ότι ε, πρόκειται για ένα πολυδιάστατο ζήτημα και πολλές φορές δεν έχουμε κατά νου τι υποστηρίζουμε συνολικά. Έχουμε μια κρίσιμη μάζα χρηματοδότησης που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά καλύτερο τρόπο. Θα πρέπει να μειώσουμε τον αρνητικό αντίκτυπο της θεώρησης του ζητήματος. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να προβάλλουμε μια στρατηγική κατά του πλαστικού σε όλους τους τομείς που προαναφέρεται. Επίσης, ε, θα πρέπει να τονίσουμε τη σημασία της Σύμβασης των ε, Ηνωμένων Εθνών για τις θάλασσες, η οποία διέπει όλες τις δραστηριότητες στον τομέα των ωκεανών και της θάλασσας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, ε, πιστεύουμε ότι θα ε, καταφέρουμε τους φιλόδοξους στόχους που έχουμε προβάλει σε αυτή τη διάσκεψη. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ήθελα ο κύριος ε, Φαρία, ο οποίος είναι εισηγητής στη δική μας έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας, να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πίτερ Τόμσον, ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Είπατε ότι σε ένα μήνα θα έχουμε τη διάσκεψη για τους ωκεανούς και οι εκπρόσωποι της ανθρωπότητας θα είναι όλοι παρόντες και το θέσατε πολύ σωστά. Τώρα, ο στόχος βιώσιμης ανάπτυξης υπαριθμών 14 θα ληφθεί υπόψη για να μην βλάπτουμε πλέον, να μην βλάπτουμε πλέον τους ωκεανούς μας. Ξέρετε ότι προέρχομαι από μία χώρα η οποία λαμβάνει πολύ σοβαρά τις κλιματικές αλλαγές. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ταχύτερο δυνατό γιατί νιώθουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη χώρα μου. Μιλήσατε για τα πλαστικά απόβλητα και τα συναφή ζητήματα, κάτι το οποίο δείχνει ότι η διεθνής κοινότητα ανησυχεί ιδιαίτερα για τις αρνητικές επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας που πλήττει τους ωκεανούς μας. Και εμείς ως ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα είμαστε παρόντες. Εγώ είμαι εισηγητής για την πρωτοβουλία για την διακυβέρνηση των ωκεανών και θα είμαι παρόν και προσμένω και τα αποτελέσματα της διάσκεψης. Υπάρχουν τόσα ερωτήματα που θα μπορούσα να σας υποβάλω, αλλά θα αρκεστώ σε δύο. Ζητήματα που με ανησυχούν ενώ Ποιες είναι οι προσδοκίες μας από τη διάσκεψη αυτή. επειδή είστε Αμερικανός, σας το θέτω. Ε, πώς μπορείτε να αποκλίνετε από την πολιτική Τραμπ σε σχέση με τις κλιματικές αλλαγές που αφορά μια παγκόσμια προσπάθεια. Επίσης μιλάμε για τη διακυβέρνηση των ωκεανών και υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο με απασχολεί ε, δηλαδή σε σχέση με τις ε, ε, εκπομπές που προκύπτουν από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες και τη μείωσή τους. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε μέσω του IMO που είναι ένας οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, τα τελευταία χρόνια δεν έχει ληφθεί υπόψη η αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος σοβαρά. Θα πρέπει και εμείς να ασχοληθούμε με ε, θέματα εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα σε σχέση με τις ναυτιλιακές δραστηριότητες. Στη χώρα μου αντιμετωπίζουμε ένα μείζον ζήτημα που αφορά την ε, διακυβέρνηση των ωκεανών σε σχέση με την ε, εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου υπερακτίως. Ο Υπουργός ε, Θαλασσίων Δραστηριοτήτων ε, βρέθηκε στη ΣΥΠΑ και είπε στην κυβέρνηση, τον είπα, ότι θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε την ε, τεχνογνωσία μας σε σχέση με τις περάκτιες δραστηριότητες και ίσως να επεκταθείτε και εκεί. Κάτι το οποίο με απασχολεί ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε κύριε Φαρία. Τώρα κύριε Τόμσεν, θα ήθελα να στραφώ σε εσά για τα σχόλιά σας. Για όλα τα σχόλια τα οποία εφήγησαν. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω ότι είμαι μεταξύ των δικών μου ανθρώπων, ανάμεσα στους δικούς μου ανθρώπους σήμερα το πρωί, ανθρώπους των ωκεανών. Πρόκειται για ένα υπαρξιακό θέμα που απασχολεί την ανθρωπότητα και είναι ύψης τη σημασία σε σχέση με το οξυγόνο που αναπνέουμε και τις πρωτεΐνες που καταναλώνουμε. Χαίρομαι που σας απασχολεί εξίσου για να δούμε τα σημεία ένας, ένα προς ένα. Συμφωνώ με αυτά που προείπε ο κύριος Γιαβόρ και πρέπει να τονίσω ότι όταν ήμουν στην Ουγγαρία νωρίτερα φέτος με ε, εξέπληξε το πόσο αντιμετωπίζει, πώς ανταποκρίνεται αυτή η χώρα στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, σε όλους τους στόχους ταξιδεύοντας ανά τον ε, κόσμο και νωρίτερα παρευρέθηκα στην Κίνα και την Ινδία και ήρθα σε επαφή με τους πρωθυπουργού και τις κυβερνήσεις και είδα ότι οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ε, της ατζέντα αυτών των χωρών με βάση τους στόχους για το 2030. Άρα μετά την Κίνα και την ε, Ινδία είδα ότι όλοι οι, οι, οι υπουργοί ανταποκρίνουν σε αυτούς τους στόχους, όπως και ο τόπος από όπου προέρχομαι, η νήσι Φίτζη δηλαδή. Και υπάρχει πλήρη συνεργασία σε αυτό το τομέα. Δυστυχώς, πολλοί μεμονωμένοι φορείς δεν κατανοούν αυτούς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Εγώ ε, ελέγχω την κατάσταση στις ε, ε, δεξιώσεις ή στα ξενοδοχεία, γιατί πολλοί δεν γνωρίζουν τι είναι οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης. Πολλές φορές μου λένε SDG, τι είναι αυτό. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν οι επιλογές, οι καθημερινές μας επιλογές παραγωγής και κατανάλωσης. Κάτι το οποίο θα πρέπει να ε, μεταβάλουμε γιατί δεν υπάρχει βιωσιμότητα αν συνεχίσουμε έτσι. Μιλάμε για μια αύξηση της ε, θερμοκρασίας κατά 3 ή 4 βαθμούς τη στιγμή που θα πρέπει να μείνουμε κάτω από τους 2 βαθμούς. Και γνωρίζετε ότι η μεσαία τάξη ε, μεγενθύνεται κατά εκθετικό τρόπο και περισσότεροι από εσά, περισσότεροι από που βρισκόσαστε στη μεσαία τάξη, ξέρετε ότι πολλές φορές, όπως και εγώ, υπερκαταναλώνουμε, θέλουμε μια δεύτερη τηλεόραση, ένα δεύτερο αυτοκίνητο. Ε, έχω έχουμε μεγάλες ανάγκες και δεν θα μετατρέψουμε, δεν θα μετασχηματίσουμε τον κόσμο εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι, αλλά οι νέοι, οι νέοι και τα παιδιά τους, γιατί θα αντιμετωπίσουν μεγάλες δυσκολίες αν δεν αλλάξουμε το σχήμα μας κατανάλωσης και παραγωγής για την Ατζέντα 2030. Η εκπρόσωπος από τη Γαλλία μίλησε για, τις υπερπόντιες, για τα υπερπόντια διαμερίσματα. Θα ήθελα να πω ότι η ατζέντα του 2030 αφορά όλους τους ωκεανούς και περιφέρειες και από επισκέψεις στα υπερπόντια διαμερίσματα είδα ότι το ίδιο ισχύει και εκεί. Ίσως τα προσωπικά σχήματα και επιλογές δεν είναι καλά. Στον εκπρόσωπο της Ιταλίας θα ήθελα να πω ότι η Ιταλία τα τελευταία δύο χρόνια έχει συνεισφέρει ιδιαίτερα ε, στην προστασία των ωκεανών. Στη Ρώμη πέρσι η επιστημονική κοινότητα και η επιχειρηματική κοινότητα συνεργάστηκε με τα Ηνωμένα Έθνη και τα εμπλεκόμενα κράτη. Και είδαμε ότι αυτή η συμβολή όλων μπορεί να ενεργοποιήσει αυτόν τον τομέα και να του δώσει μια νέα δυναμική, συμμετοχική δυναμική και η Ιταλία μαζί με το Παλάου αυτή τη στιγμή ε, έχει αναλάβει την προεδρία ενός από αυτούς τους, από αυτούς τους ε, διαλόγους στους οποίους προαναφέρθηκα. Όταν μιλάμε για γαλάζια ανάπτυξη μιλούμε περισσότερο για ε, γαλάζια οικονομία. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει λέξη βιώσιμη και ε, μπροστά στην ανάπτυξη και μπροστά στην οικονομία. Εγώ ασχολήθηκα ε, με αυτό το θέμα όλη μου τη ζωή, αρχίζοντας το 72 μετά από το ε, πτυχίο μου από το Cambridge και ειδικεύτηκα σε αυτόν τον τομέα και είδα ότι πολλοί άνθρωποι βρίσκονται στα όρια της ε, ένδυας, ιδιαίτερα σε παραγκουπόλεις εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων ή στις αγροτικές περιοχές και τώρα είμαι πεπισμένος ότι μπορούμε να προωθήσουμε βιώσιμους στόχους και βιώσιμη ανάπτυξη. Βρισκόμαστε στη σωστή οδό πλέον. Στην εκπρόσωπο της ε, Γερμανίας, την κυρία... Α, με συγχωρείτε, στην αυστριακή εκπρόσωπο, την κυρία Κάντενμπαχ, ε, ε, το HOPF, το πολιτικό φόρουμ υψηλού επίπεδου, είναι αυτό που αναλαμβάνει αυτό τον συντονισμό. Και φέτος 40 χώρες θα παρήσανται τον Ιούλιο για να μας πούν τι κάνουν σε σχέση με τους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι μια χιονοστιβάδα και θα πρέπει να προβάλλονται οι καλές ιδέες από όλες τις χώρες να δούμε πού επιτυγχάνουμε, πού αποτυγχάνουμε και ούτω καθεξής. Ως προς την κυρία Μάισνερ, μίλησε για βιώσιμη γαλάζια ανάπτυξη. Στο Woods Hole, στο Οκεανογραφικό κέντρο στις, στη Μασαχουσέτη, α, κυρία Μάισερ, τώρα σας, βλέπω, βλέπουμε ότι αυτό το Οκεανογραφικό Ινστιτούτο είναι από τα μεγαλύτερα μετά από τη Γαλλία και τη Βραζιλία προβάλλονται τα ε, μεγαλύτερα αιτήματα από, το, από αυτό το ωκεανογραφικό κέντρο. Γιατί στην ουσία στο μέσο του ωκεανού τι κάνουν, ε, καταγράφουν τα πλανκτόν και βλέπουμε τις μικρομορφές ζωής που τρώνε το μικροπλαστικό. Και αυτό είναι φοβερό να το βλέπει κανείς ε, ε, σε φιλμ. Δηλαδή βλέπουμε ε, τι γίνεται. Τα μικρά ψάρια τρώνε το πλαστικό, μετά τα τρώνε τα μεγάλα ψάρια και καταλήγουν στο τραπέζι σας και στην ουσία τρώτε πλαστικό. Άρα στη διάσκεψη θα βασιστούμε σε επιστημονικά δεδομένα και αυτές οι εταιρικές σχέσεις και ο διάλογος αφορά την αντιμετώπιση της μόλυνσης σε επιμέρους τομείς. Έχουμε συγκεκριμένους οργανισμούς που μας λένε τι συμβαίνει, μας λένε την αλήθεια. Δεν πρόκειται για εικασίες. Και μετά βλέπουμε πώς μπορούμε να επιλύσουμε τα ζήτηματα αυτά. Εάν βρούμε καλές λύσεις, τότε θα πρέπει εκεί να προβληθούν γιατί ε, από τον εταιρικό αυτό διάλογο θα βρεθούν οι καλύτερες λύσεις σε περιβαλλοντικό επίπεδο και μιλώ για όλους, για την ανθρωπότητα. Δεν πρόκειται για ιδιοκτησία ορισμένων γραφειοκρατών των είπα μιλήσατε για τις... για τις ε, εξορίξεις στο βυθό της θάλασσας. Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τι γίνεται. Το είδαμε αυτό και στη, στα Φίτζη και θεωρούμε ότι η εξορίξη στην ε, υφαλοκρηπίδα είναι κάτι το πολύ ε, σημαντικό στη χώρα μου, στις νήσους ε, Φίτζη. Είμαστε οι πρώτοι που υπογράψαμε αυτή τη σύμβαση. Τώρα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η εξορίξη στο βυθό της θάλασσας αποτελεί, αποτελούν πραγματικότητα. Δεν ξέρουμε πώς θα γίνει και πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το ε, θέμα ο Διεθνής Οργανισμός Υφαλοκρηπίδας, αλλά προωθούμε τον νόμο για να δούμε πώς μπορούμε να ε, έχουμε μια διαδικασία πιστοποίησης και αδειοδότησης για τις εξορίξεις αυτές. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι η υφαλοκρηπίδα που καλύπτει το 50% των ωκεανών ε, αποτελεί εγγύηση γιατί Κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς ε, προέγκριση. Άρα αυτό είναι καθησυχαστικό. Το BBNJ, δηλαδή η βιοπικιλότητα πέρα από την εθνική δικαιοδοσία, η BBNJ, μας αρέσουν τα ακρόνιμά μας, ε, μας απασχολεί ιδιαίτερα η Βραζιλία είναι πρόεδρος και στην ουσία τι γίνεται, η πειρατεία ισχύει πάνω από την ε, ε υφαλοκρηπίδα και μέχρι την ίσαλογραμμή. Και νομίζω ότι έτσι θα πρέπει να ασχοληθούμε με τη ε, θάλασσα. Είναι η κοινή μας κληρονομιά. Άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ υπεύθυνοι μέσα στα πλαίσια αυτού του φορέα, του BB&J. Η Πορτογαλία έχει επιτελέσει μεγάλο έργο μέσα στα πλαίσια της διαχείρισης των ωκεανών. και χτες αφού συναντήθηκα με τον Επίτροπο Βέλα ε, μιλήσαμε για τη συμμετοχή αυτή στο, στη διάσκεψη των ωκεανών και το θέμα των εξοπλισμών είναι ύψης της σημασίας και χαίρομαι που και ο κύριος Βέλα θα παρευρεθεί στη διάσκεψη. Σε σχέση με τη διάσκεψη των ωκεανών, είπα στον κύριο Βέλα ότι το, ο, ο στόχος βιώσιμης ανάπτυξης παριθμών 14 είναι το μόνο μέσο για να ε, μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την υγεία των ωκεανών. Έχουμε και το θέμα του ειρηνικού με την αλίευση τόνου και ούτω καθεξής. Είναι πολύ καλές ε, αυτές οι πρωτοβουλίες και τις υποστηρίζουμε μέσα στα πλαίσια του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης παριθμών 14, αλλά παγκοσμίω υπάρχει μόνο η διάσκεψη των ωκεανών, η οποία θα λάβει χώρα τον Ιούνιο στις ΗΠΑ και θα συνεχίσει αυτή την ε, παγκόσμια προσπάθεια μέχρι το 2030, γιατί αυτή είναι η εντολή μας. Νομίζω ότι κάλυψα όλα τα σημεία. Α, κύριε Φαρία. Ο κύριος Φαρία υπέβαλε δύο ερωτήσεις για τη θέση των ΗΠΑ της κυβέρνησης. Ε, μην προτρέχετε αφήστε να καταλαγιάσουν τα πράγματα, δεν υπάρχει ακόμα σαφής πολιτική. Για τους ωκεανούς ε, βρισκόμαστε σε μία μεταβατική περίοδο ακόμα. Σε σχέση με τις εκπομπές από τον, τον τομέα της ναυτιλίας, έχουμε ασχοληθεί μαζί με τον ε, ΠΟΕ για το αντι και τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και θα μας απασχολήσει το θέμα και στη διάσκεψη των ωκεανών. Για τη διάσκεψη των ωκεανών θα ήθελα τελικά να πω ότι έχει γίνει μεγάλη εργασία τα τελευταία δύο χρόνια σε καθημερινή βάση και είμαι πεπισμένος ότι αυτή θα είναι η αλλαγή που αποζητάμε είμαι πεπισμένος ότι θα φτάσουμε στους στόχους μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακροασή σας. And, uh, inspiring on our work. Good luck with the conference. We will all try to support this initiative and I have towards sustainable growth. Thank you. Thank you very much. Good morning, everyone. I invite you to take your seats, prepare your uh, voting cards. Σας παρακαλώ πολύ ε, να λάβετε την ε, κάρτα σας για να ψηφίσετε. Δεν είναι δύσκολη η ψηφορία μας. Έχουμε δύο-τρεις ε, ψηφορίες. Λοιπόν, πρώτη ψηφοφορία. Ε, τρεις ε, ψηφοφορίες έχουμε για αντιρρήσεις ε, με βάση τον κανόνα 106. Πρώτα θα ψηφίσουμε για την αντίρρηση σχετικά με το γενετικά τροποποιημένο βαμβάκι. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η κυρία Γκαρντίνη. Δυστυχώς δεν ακούμε εμείς, είναι κλειστό το μικρόφωνο της. Θα το λάβουμε υπόψη μας ε, και θα αλλάξουμε την ψήφο σας, ε, το πώς ψηφίσατε. Επόμενο θέμα, αντίρρηση για τροποποιημένο ε, αραβόσιτο. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και τελευταία ψηφοφορία, πάλι μια αντίρρηση για τις ε, βέλτιστες ε, διαθέσιμες τεχνικές για μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν ολοκληρώσαμε τις ε, ψηφοφορίες για σήμερα. Να κάνουμε σύντομο διάλειμμα. So, dear colleagues, we... I propose you to start the next uh, item on the agenda. Ε, να ξεκινήσουμε το επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη, ε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, είναι το σχέδιο έκθεση για τον περιορισμό τη χρήση κάποιων επικίνδυνων ουσιών στο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Είμαι επικεφαλής και υπεύθυνη της ε, έκθεσης αυτής. Το ζήτησαν οι συντονιστέ. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, λοιπόν, να σα πω δύο λόγια για την έκθεση αυτή. Καλωσορίζω την νομοθετική πρόταση της Κομισιόν που είναι απαραίτητο βήμα για να επιληθεί το πιεστικό πρόβλημα που συνδέεται με την τρέχουσα διατύπωση της ΡΟΣ 2 ε, για να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου διατηρώντας το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Για αυτό το λόγο προσπαθούμε να προχωρήσουμε γρήγορα σε αυτό το φάκελο. Η αναθεώρηση του πεδίου εφαρμογής της ΡΟΣ 2 θα εξασφαλίσει ή θα διατηρήσει τις θέσεις απασχόλησης στι μικρέ και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα υποστηρίξει τον τομέα της δημόσια υγείας, γιατί θα έχουμε ένα ανανεωμένο, ανακαινισμένο ε, ιατρικό εξοπλισμό και θα προωθήσει την κυκλική οικονομία. Ο στόχο τη ε, επανεξέτασης αυτής του πεδίου δεν είναι να εξεταστεί ολόκληρη λειτουργία τη ε, ΡΟΣ 2, πιστεύω ότι οι πιθανές βαθύτερες αλλαγές στην οδηγία αυτή δεν θα πρέπει να είναι ο σκοπός αυτής της διαδικασίας, αλλά αντίθετα ο σκοπός της επικείμενης γενικής αναθεώρησης της οδηγίας που θα διενεργηθεί από την Επιτροπή έως τις 22 Ιουλίου του 2021, όπως ορίζεται στην ε, οδηγία. Όμως η επανεξέταση αυτή του πεδίου εφαρμογής αποτελεί ευκαιρία για να δούμε κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της γενικής αναθεώρησης. Με, αυτή ε, με αυτό το σκεπτισμό ε, ε, η, το σχέδιο έκθεσης αφορά ε, τα εξή θέματα. Θα πρέπει η επερχόμενη αναθεώρηση να συνοδεύεται από ε, νομοθετική ε, πρόταση με σαφή μεθοδολογία για όλα τα βήματα που οδηγούν στην τροποποίηση του καταλόγου των ε, ουσιών υπό περιορισμό και των ε, εξαιρέσεων. Θα πρέπει να υπάρχει γνωμοδότηση της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για τα Χημικά, μια και έχουμε αυτή την υπηρεσία, γιατί να μην τη χρησιμοποιήσουμε. Και ένα άλλο θέμα είναι, λόγω του αυξανόμενου αριθμού εξαιρέσεων και περιπλοκών της οδηγίας για να υπάρχει και προκλεψιμότητα και ασφάλεια δικαίου, μια νέα ε, ανάγκη η Κομισιόν να μας δίνει ξεκάθαρο ε, χρονοδιάγραμμα για την υιοθέτηση της απόφασής της ένα μήνα μετά την ε, λήψη της οποιασδήποτε αίτηση για εξαίρεση. Ε, επίσης, θα πρέπει να πλουστευτεί η διαδικασία για τις ε, κατεξιόδηση πράξεις, για τις εξαιρέσεις, για να καλυφθούν περιορισμένα τεχνικά θέματα Αυτό πρέπει να προσθεθεί. Αυτά με δύο λόγια είναι η ουσία αυτής της έκθεσης. Τώρα θα ήθελα να καλέσω τους σκιώδεις εισηγητές να δώσουν τη γνώμη τους. Και ο πρώτος είναι η κυρία Κάντεμπεργκ. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την ε, Πρόεδρό μας ε, που παράλληλα είναι και η σε αυτό το θέμα. Νομίζω οι περισσότερες ε, προτάσεις ε, που θέλω να κάνω για να συμπληρώσω αυτά που ακούστηκαν, οι περισσότερες ε, είναι με θετικό πρόσημο. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι στο τέλος Βιγάκη, εκεί που μιλήσατε για την μελλοντική πρόσβαση, αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει είναι στη διαδικασία της συναπόφασης που έχουμε να υπάρχει επιπρόσθετα και η δυνατότητα σε όλους τους τομείς να προσθετούν συγκεκριμένες μέθοδοι. Νομίζω ε, στην περίπτωση αυτή, αν προέκυπτε κάτι τέτοιο, θα οδηγούσε σε καθυστέρηση των συγκεκριμένων βημάτων και επίσης ε, θα οδηγούσε στο να ε, δοθεί υπερβολική σημασία στη βιομηχανία. Θα έχει άποψη η βιομηχανία και κατά την άποψή μου αυτό θα οδηγούσε σε ατέρμονους ε, αγώνες και διενέξεις επί της ουσίας Πρόκειται συγκεκριμένα για τις τροπολογίες 4 και 5, για αυτές τις δύο τροπολογίες. Εγώ προτείνω να μην στηριχτούν αυτές οι δύο τροπολογίες. Και όπως είπε και η προλαλήσασα, η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι καλή, οδηγεί στο στόχο, ε, μόνο που εμείς πιστεύουμε ότι θα έπρεπε ήδη να έχει κατατεθεί από το 2014. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για τη δουλειά που μας έκανε, λέει ο κύριος Σουίτεμα. Όπως εξηγήσατε, κάποιες κατηγορίες ηλεκτρονικού εξοπλισμού, χωρίς να το θέλουμε, θα απαγορευτούν από την ε, δευτερογενή αγορά ε, στις 22 Ιουλίου, από τις 22 Ιουλίου του 2018 και μετά. Δεν είναι σωστό αυτό. Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα είναι η δυνατότητα να χρησιμοποιούμε τα ανταλλακτικά. Εάν δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα ανταλλακτικά, κάποιε από τις συσκευέ δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν πια. Ακόμα και αν θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν πολύ, να έχουν χρόνο ζωή μπροστά του. Αυτά τα δύο παραδείγματα δείχνει ότι αυτό, αυτή η οδηγία είναι κατά του στόχου της κυκλικής οικονομίας και θα δημιουργήσει και οικονομικές ζημίες για τους ε, κατόχους και παραγωγούς ε, αυτών των ε, προϊόντων με μεγάλο κύκλο ζωής. Γι' αυτό λοιπόν καλωσορίζω την πρόταση της Κομισιόν και καλωσορίζω την προσθήκη σας. την προσθήκη που κάνατε τη πρόταση τη Κομισιόν στη δική σα έκθεση. Όμω, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μπαίνουμε σε υπερβολικέ λεπτομέρειε για πιθανέ νομοθετικέ προτάσεις το 2021. Ε, κύριε Κλόνεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ κύριε Συγκήτρια, Πρόεδρε και Συγκήτρια δηλαδή. Θαυμάσια η δουλειά σας. Και εγώ υποστηρίζω απόλυτα το μήνυμα της ΕΚΑ Και εγώ έχω να κάνω κάποιες τροπολογίες σε σχέση με τον ηλεκτρικό εξοπλισμό που ανακαινίζεται εκ των υστέρων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας ότι με την ε, εκτονιστέρων των ανακαίνιση του υπάρχοντος εξοπλισμού και την αναβάθμισή του, ας πούμε, μπορούμε να του δώσουμε μεγαλύτερο κύκλο ζωής, εν πάση περιπτώσει, να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία που εμπεριέχεται σε αυτές τις συσκευέ. Ευχαριστώ από τους πράσινους. Ποιος είναι? Η κυρία Ντορνάνου. Ευχαριστώ. Καταρχά, να σε ευχαριστήσω Πρόεδρε για τη δουλειά που κάνατε, πολύ ποιοτική για αυτό το τεχνικό θέμα, καθώς και για τις ε, διευκρίνήσει ε, που υπάρχουν στο σχέδιο εκθεσή σας. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ε, που αφορά την πλαισίωση και τον περιορισμό της χρήση κάποιων ουσιών επικίνδυνων στις, στο, στα ηλεκτρικά στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό θα πρέπει να έχει σαν στόχο τη μείωση του κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Πρώτο στόχο πρέπει να είναι αυτό. Συμφωνώ με την ανάγκη λοιπόν να δούμε τι παρενέργειε τη οδηγία του 2011 στα πλαίσια μια πραγματική κυκλική οικονομία. Όμω, είναι πολύ σημαντικό αυτή η προσέγγιση να σεβαστεί την αρχή της αναλογικότητας και της επικουρικότητας ε, που εγγυάται η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνώ με αυτό που είπε η συγκήτρια ε, για τις βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν τη δράση μας πολύ περισσότερο παραποτέ θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την, ε, το σωστό βίο και κύκλο ζωή στι ε, ηλεκτρικέ και ηλεκτρονικέ συσκευέ και θα καταθέσω και σχετικέ τροπολογίε. Σε ό,τι αφορά τι νέε αιτήσει για ανακαίνιση ή εξαιρέσει, αυτοί οι έξι μήνε που αφήνουμε στην Κομισιόν για να δράσει, συμφωνώ με τι ειδικέ περιπτώσει που μπορεί να δικαιολογούν μια επιπλέον ε, καθυστέρηση. Όμω, εάν θέλουμε να έχουμε δίκιο ανταγωνισμό στον τομέα που, στους τομείς που χρησιμοποιούν επικίνδυνες ουσίες στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό είναι σημαντικό να δώσουμε στις επιχειρήσεις ένα νομικό πλαίσιο ασφαλές ούτω ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι αυτής της οδηγίας. Σας ευχαριστώ. Ποιος θέλει άλλο στο λόγο. Ο, ε, ο, διευθυντής, ε, ο αρπόδιος διευθυντής της Κομισιόν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ που οργανώνετε αυτή τη συζήτηση, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και για την έκθεσή σας. Κάναμε μια πρόταση, λίγο καθυστερημένα, σωστό είναι από ό,τι σχεδιάζαμε αρχικά, για την τροποποίηση αυτής της οδηγίας, αλλά το κάναμε μαζί μαζί με την έκθεση για το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία. Υπάρχει λόγος. Γιατί οι τροπολογίες δεν είναι τα τμήμα του σχεδίου δράσης. Γιατί οι τροπολογίες ακολουθούν τη λογική της κυκλικής οικονομίας και ο ορισμός της κυκλικής οικονομίας είναι να ε, διατηρήσουμε την αξία των υλικών και εξοπλισμών το συντομότερο όσο περισσότερο γίνεται. Η τροπολογία ακριβώς αυτό το λόγο εξυπηρετεί ανταποκρίνεται σε ένα αίτημα ε, για την αναθεώρηση του πεδίου και την επανεξέταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, ε, αλλά μην ξεχνάτε και ότι κάναμε και πολύ περίπλοκες ε, διαβουλεύσεις με τους ενδιαφέρομενου φορείς και μια μελέτη αντικτύπου. Κάναμε δηλαδή ανάλυση του τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή τη φάση και ακριβώς αυτό προτείνουμε. Οι αλλαγές θα διευκολύνουν ε, τις ε, επιχειρήσεις στη δευτερογενή αγορά, την μεταπόληση ας πούμε και την μετασκευή και διόρθωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και θα ε, εξοικονομήσει δημόσιο χρήμα και θα διατηρήσει τους δημόσιους πόρους. Επίσης έχουμε δύο περιορισμένες αποκλεισμούς από το πεδίο της ΡΟΣ, κυρίως για τα εκκλησιαστικά όργανα, για λόγους πολιτιστικής κληρονομιάς ε, και, κάποιους ε, και κάποια μειωδικά ε, κινητά μηχανήματα. Δεν θα μειώσει αυτό την προστασία του περιβάλλοντος. Πιστεύουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία για την επανεξέταση του πεδίου εφαρμογή της ΡΟΣ ε, θα μπορούσε να κλείσει γρήγορα μέσω σοβαρές θετικές περιβαλλοντικές και οικονομικές συνέπειες. χωρίς να προδικάσω τελική θέση της Κομισιόν, Παραδείγματο χάρη μπορεί να συνδυάσουμε διάφορες ε, τεχνικέ ε, συναφεί αποφάσεις σε μία ε, κατεξιοδότηση πράξη. Μπορεί αυτό να διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων υπό την οδηγία. Επίσης, καταλαβαίνω ότι έχετε πρόβλημα με την αδυναμία μας συχνά να σεβαστούμε τους έξι μήνες, συχνά για αντικειμενικούς λόγους, επειδή πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιες διαδικασίες, νομικές διαδικασίες. Δεν μπορούμε να σεβαστούμε αυτές τις, αυτό το εξάμεινο, όπως παραδείγματος χάρη δημόσιες διαβουλεύσεις, ας πούμε, που κρατάνε ένα-δύο μήνες. Ε, και επίσης η περίοδος ε, αντίρρησης ή μη αντίρρησης από, τα, από τους φορείς. Επίσης ε, δύο μήνες που θα πρέπει να κάνουμε κοινοποίησει, μεταφράσει μετά. Ε, σοβαρή ανάλυση και συνήθως το κάνουμε αυτό μέσω εξωτερικών συμφούλων ε, που πρέπει να σεβαστούν το ε, συμβατικό δίκαιο, συχνά όλο αυτό περιμέ... Ε, μας παίρνει 24 μήνες. Ε, επομένως, πώς να σεβαστούμε το εξάμεινο. Ε, Καλωσορίσω λοιπόν την πρότασή σας. Να ξεχάσουμε αυτή την προθεσμία. Υποστηρίζω όμως την ιδέα που εκφράσετε να δώσουμε εμείς ένα χρονοδιάγραμμα στους ενδιαφερόμενους φορείς, που δεν θα είναι όμως και αμετάβλητο, έτσι. Θα, λέμε έτσι χοντρικά ότι γενικά για τις εξαιρέσεις αυτό το χρόνο χρειαζόμαστε για να εξετάσουμε και να διεκπαιρεώσουμε την αίτηση εξαίρεσης. Νομίζω ότι αυτό τους δίνει μια ασφάλεια δικαίου. Επίσης η υπηρεσία ΕΚΑ ε, θα μπορούσε να ε, συνεισφέρει και αυτή στην ε, σύνταξη των κατεξιοδότηση πράξεων Πιστεύουμε ότι η ΕΚΑ τώρα έχει τη γνώση, την καλύτερη γνώση στον κόσμο για χημικές ουσίες, επομένως κάποια στιγμή πρέπει να βασιστούμε στη γνώμη της. Το θέμα είναι το κάνουμε τώρα ή ε, θα τα κάνουμε στα πλαίσια της γενικότερης επαναθεώρησης ε, που θα γίνει μετά από κανένα δύο χρόνια όταν θα έχουμε ξαναεξετάσει όλες τις δυνατότητες. Πάντως, έχει νόημα να προσφύγουμε στην ΕΚΑ και υποστηρίζω αυτή την ιδέα χωρί βεβαίω να προδικάσω την τελική θέση τη Κομισιόν. Επίση, το δικαίωμα πρωτοβουλία τη Κομισιόν θα πρέπει να διατηρηθεί, μην το ξεχνάμε αυτό, και οι τροπολογίε σε ό,τι αφορά το μέλλον της πρότασης, όταν είναι επιτακτικέ είναι προβληματικέ. Η ιδέα τη διευκρίνηση των μεθοδολογιών, όταν είναι ειδικά επιτακτικέ και ότι θα πρέπει να κάνουμε κάτι στις ε, μελλοντικέ τροπολογίε, αυτό προδικάζει τις ε, επακόλουθες ε, τροπολογίες. Το θέμα είναι βεβαίως να, ε, να αξιολογούμε τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε για την προσθήκη ουσιών. Αυτό ναι, έχει νόημα. Όμως τα μεγαλύτερα θέματα θα πρέπει να τα αφήσουμε για αργότερα. Μετά από κάνα δύο χρόνια που θα κάνουμε πλήρη μελέτη αντικτύπου, πλήρη δημόσια διαβούλευση και αυτό θα χρειαστεί χρόνο όπως καταλαβαίνετε. αλλά πρέπει να επιλύσουμε τα θέματα που προβλέπονται προς επίλυση στην ε, επερχόμενη αναθεώρηση. Σας ευχαριστώ που συμφωνείτε και θα συμφωνήσετε ταχύτερα σε αυτή την πρόταση, που νομίζω ότι είναι μια πρόταση κοινή λογικής. Έτσι θα την ονόμαζα. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ και εγώ για την, ε, για την παρέμβασή σας. Νομίζω ότι υπάρχει απόλυτη σαφήνεια τώρα και διαφάνεια. Δεν προδικάζουμε τίποτα επίσης και νομίζω βοηθάμε και τον κλάδο. Και εμείς εργαζόμαστε με τον ε, ενδεδειγμένο τρόπο. Αυτή ήταν, ε, αυτός ήταν ακριβώς ο σκοπός αυτής της προσπάθειας, αυτού του εγχειρήματο να υπάρξει σαφήνεια. Δεν υπάρχει τίποτα επιτακτικό εδώ, απλώς ενδείξεις δίνουμε για το τι θα θέλαμε να δούμε στο μέλλον, στη μελλοντική αναθεώρηση. Έχουμε χρόνο μέχρι την αναθεώρηση. Να βελτιώσουμε τον τρόπο εργασίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή. Έχουμε μία προθεσμία για τις τροπολογίες που είναι η αυριανή ημέρα. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών ε, αύριο 12 η ώρα. 11 ε, η ώρα, συγγνώμη, και ψηφίζουμε στην Επιτροπή στις 13 Μαΐου. 13 Μαΐου. Σας ευχαριστώ πολύ. Το επόμενο σημείο είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον εκτελεστικό διευθυντή της ΕΦΣΑ. Αλλά έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα μέχρι τις 11 παρατέταρτο ας πούμε. Έτσι, 5 λεπτά και κάτι διάλειμμα. So, um, I think we can resume the work. Um, I want to say hello to the Executive Director of the European Food Safety Authority, Dr. Bernard Url. Λόγο έχει ο κύριος Ουρλ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. και θα μιλήσουμε για την ε, πορεία της ΕΦΣΑ το 2017-19. Ο δόκτωρ Ούρλ θα λάβει το λόγο για να μας παρουσιάσει και το ετήσιο πρόγραμμα και όλες τις εξελίξεις. Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα σας και από τη δική μου πλευρά. Είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι εδώ και να συζητώ μαζί σας. Δεν είναι εύκολο, αλλά προσωπικά το ευχαριστιέμαι να προβούμε σε ανταλλαγή απόψεων για την ασφάλεια τροφίμων. Επίσης θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξή σας κατά την διαδικασία της απαλλαγής Και σας ευχαριστώ γιατί την προηγούμενη ε, εβδομάδα αναλάβατε αυτή την πρωτοβουλία για την προστιθέμενη αξία των ε, ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για τη δημόσια υγεία. Συνεργαστήκαμε και με άλλους οργανισμούς επί του θέματος. Θα ήθελα στην εισήγησή μου να ασχοληθώ με ορισμένες προκλήσεις για την ΕΦΣΑ γιατί είναι θέματα που θα ανακύψουν και κατά τη συζήτηση. Θα πρέπει όμως να πούμε ότι η ΕΦΣΑ χάρη στην υποστήριξη των ε, εμπειρογνωμών των κρατών μελών, ένας μικρός οργανισμός ε, διεθνός έχει καταφέρει να δώσει πολύ καλό ποσοτικό και ποιοτικό output. Βρέθηκα στην ε, Ιαπωνία την προηγούμενη εβδομάδα με την ομάδα αξιολόγησης της ε, Γερμανίας και της Γαλλίας και το πρότυπο της ΕΦΣΑ εκτιμήθηκε στην Ιαπωνία και στην περιοχή ΑΖΕΑΝ και χαιρόμαστε ότι το πρότυπο που δημιούργησε το Κοινοβούλιο το 2002 με 80 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, έδωσε ε, χιλιάδες επιστημονικών output και φτάσαμε και σε παγκόσμια ε, επίπεδα και πρότυπα αξιολόγησης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα, τις οργανώσεις των κρατών μελών και τους εμπειρογνώμονες που μας βοήθησαν να τα καταφέρουμε γιατί εργαζόμαστε με εθελοντές, εμπειρογνώμονες των κρατών μελών που είναι εθελοντές για το ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα. Και εάν συνεργαζόμαστε ε, είναι πραγματικά εκπληκτική η διάθεσή τους, η καλή διάθεση συνεργασίας και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω και τα κράτη-μέλη γιατί επιτρέπουν στους εμπειρογνώμονες να συνεργαστούν με την ΕΦΣΑ. Και θα ήθελα τώρα να ασχοληθώ με αυτή την πρώτη πρόκληση. Πώς τα κράτη-μέλη και στο μέλλον θα επιτρέπουν στους καλύτερους εμπειρογνώμονες και επιστήμονες να συνεργαστούν μαζί μας για 50 ημέρες. Και αυτά είναι τα όρια του συστήματος. Θα πρέπει να πληρώνουμε αυτούς τους εθνικούς οργανισμούς για να μας επιτρέπουν να απασχολήσουμε τους εμπειρογνώμονες. Άρα μιλάμε και για ένα θέμα προϋπολογισμού και ίσως θα πρέπει το Κοινοβούλιο να ξανασκεφτεί το ζήτημα. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ε, τεχνογνωσία των επιστημόνων. Το δεύτερο θέμα που ανακύπτει και από τις συζητήσεις είναι η διαφάνεια θέλουμε να είμαστε όσο δυνατόν, όσο το δυνατόν διαφανέστεροι, να λογοδοτούμε και να μας ελέγχει η επιστημονική κοινότητα. Γι' αυτό αυτό έχει σημασία και μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής μας 2020. Προσπαθούμε λοιπόν να προβαίνουμε και σε αξιολογήσεις κινδύνου. Υπάρχουν 30 μέτρα και ένα από τα αποτελέσματα είναι ότι ότι όταν ασχολούμαστε με αλλεργιογόνες ουσίες τους γενετικούς τροποποιημένους οργανισμούς, συνεργαζόμαστε και με τους εμπλεκόμενους φορείς μέσα στα πλαίσια ε, όλου του κύκλου ζωής των προϊόντων. Αυτή είναι η διαφάνεια της διαδικασίας. Ως προς την διαφάνεια επιστημονικών στοιχείων, εμείς προσπαθούμε να ε, δώσουμε αυτά τα στοιχεία, να τα χορηγήσουμε δημοσίως, να διαδοθούν αυτά τα στοιχεία και η κοινωνία των πολιτών είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένη. Υπάρχει όμως το θέμα των ε, συγκεκριμένων μελετών του επιστημονικού κόσμου των βιομηχανιών. Στην περίπτωση της γλυφοσάτης έχουμε δημοσιεύσει 6.000 σελίδες συνοψίσεων στην ιστοσελίδα μας. Άρα η διαφάνεια είναι τεράστια ως προς την χρήση δεδομένων και προσπαθούμε να αυξήσουμε αυτή την διαφάνεια. Αλλά φυσικά υπάρχει μεγάλη πίεση και ένταση μεταξύ πλήρους διαφάνειας και του δικαιώματος προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό δεν είναι επιστημονικό ζήτημα. Υπάρχουν όρια για την ΕΦΣΑ. Δηλαδή έχουμε δώσει 10.000 σελίδες για τη γλυφοσάτη σε ευρωβουλευτές που ζήτησαν αυτά τα στοιχεία έτσι ώστε να γίνει μια νέα αποτίμηση κινδύνου της γλυφοσάτης και να δούμε πώς ορίζονται αυτά τα στοιχεία. Γι' αυτό νομίζω ότι φτάσαμε στα όρια μας και μπορεί να μας μιλήσει η βιομηχανία γιατί δίδουμε πολλά στοιχεία ή η ΜΚΟ που μας λένε ότι δεν είμαστε όσο διαφανείς θα έπρεπε αλλά εδώ είναι πολιτική απόφαση, όχι επιστημονική. Δεν είναι επιστημονικό το θέμα πόσο μακριά μπορούμε να προχωρήσουμε στη διαφάνεια. Εσείς θα αποφασίσετε κατά πόσο χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια. Και αν χρειάζεται θα πρέπει να γίνει μια νέα νομοθέτηση. Οπότε η ΕΦΣΑ πρέπει να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της βιομηχανίας αλλά πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε αυτά τα στοιχεία, τα στοιχεία που προέρχονται από τη βιομηχανία, γιατί εδώ υπάρχουν ειδικά συμφέροντα. Εδώ έχουμε τις ε, κατευθυντήριες γραμμές του ΟΣΑ και τα εργαστήρια ε, είναι κατά κάποιο τρόπο ελεγχόμενα από τα κράτη-μέλη. Και εμείς επεξεργαζόμαστε την πρώτη αυτή ύλη. Δεν συμφωνούμε με τη βιομηχανία. Επεξεργαζόμαστε αυτά τα στοιχεία και μπορούμε να φτάσουμε και σε άλλα συμπεράσματα. Χρησιμοποιούμε την πρώτη ύλη, τα πρωτογενή στοιχεία, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να φτάσουμε και σε άλλα συμπεράσματα. Και επίσης ελέγχθη, η ΕΦΣΑ δεν μπορεί να διενεργήσει αυτές τις έρευνες ανεξάρτητα. Εδώ θα πρέπει να το δούμε σοβαρά, γιατί μιλάμε για 10.000 μελέτες ετησίως. Είναι αδύνατο να διενεργήσουμε 10.000 ε, μελέτες. Θα ήταν ασύμφορο και οικονομικά και από πλευράς ε, ζωικής ευημερίας. Άρα μιλάμε για ένα ποιοτικό έλεγχο και ο έλεγχος αυτός θα μπορούσε να ενισχυθεί σε επίπεδο κρατών μελών, δηλαδή τα πρωτογενή στοιχεία να είναι ποιοτικά. Τέλος, θα ήθελα να μιλήσω για την αυτονομία μας, αυτή την πρόκληση οι επιστημονικές αξίες βρίσκονται στο DNA της ΕΦΣΑ. Αυτός ήταν και ο λόγος σύστασης της ΕΦΣΑ, δηλαδή η επιστήμη να μείνει εκτός πολιτικής οικονομίας και λόμπινγκ. Αλλά είναι και δύσκολο το ζήτημα, γιατί όταν μιλάμε για ανεξαρτησία, φυσικά η ΕΦΣΑ δεν μπορεί να είναι 100% ανεξάρτητη σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί εσείς είσαστε η αρχή του προϋπολογισμού. Το ίδιο αφορά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ο πελάτης της ΕΦΣΑ και το ίδιο αφορά και το προσωπικό Υπάρχουν λοιπόν δεσμεύσεις, δεν μπορεί να υπάρξει 100% ανεξαρτησία, αλλά προστατεύουμε την ανεξαρτησία μας έτσι ώστε να έχουμε μία αμερόληπτη προσέγγιση επιστημονικών δεδομένων και την προστασία τους, έτσι ώστε και εσείς να εμπιστευτείτε την ΕΦΣΑ γιατί και εσείς μας είπατε πώς να σας εμπιστευτούμε εάν υπάρχουν αποκλίνουσες γνώμες. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα σύστημα ποιοτικού ελέγχου το οποίο πιστοποιείται σύμφωνα με το ISO 9000. Ε, έχουμε 21 εμπειρογνώμονες που συναποφασίσουν. Δεν αποφασίζει ένας εμπειρογνώμονας και δεν υπάρχει μεροληψία συλλέγουμε και προωθούμε την πληροφορία και χρησιμοποιούμε διεθνείς μεθόδους οι οποίες είναι διαθέσιμες και διαθέτουμε όλα αυτά τα πρότυπα στον ιστότοπό μας και αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει μία μέθοδος αριστείας έτσι ώστε να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Θέλουμε εμπειρογνώμονες που πραγματικά ενδιαφέρονται γιατί επιτελούν πολύ σημαντική εργασία στην πραγματική τους επιστημονική ζωή και θέλουμε να αποφύγουμε την σύγκρουση συμφερόντων. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας υποστηρίζει διάφορες ΜΚΟ και έχουμε ένα συνεκτικό σύστημα για να προωθήσουμε ε, ένα σύστημα ώστε να μην υπάρχει σύγκρουση δεδομένων. Τι μπορεί να προσφέρει η ΕΦΣΑ στην ε, κοινωνία της Ευρώπης. Ε, να είναι ένας επιστημονικός κόμβος που να συνδέει την κοινότητα αποτίμησης κινδύνου και να συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη και τους διεθνούς εταίρους με έναν και μόνο στόχο. Να υπάρχει πραγματική επιστημονική ανάλυση για ασφαλή τρόφιμα. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Uh, Στο, το Διευθυντή. Να ξεκινήσουμε με το σημείο επαφής. Ο... Θα μιλήσει πρώτη, κυρία Αίσου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία δηλαδή. Ήμουνα σε άλλη συνεδρίαση, γι' αυτό καθυστέρησα. Άκουσα μόνο το τέλος της ομιλίας του Διευθυντή της ΕΦΣΑ. Και το πρώτο που θέλω να πω είναι τον ευχαριστώ για την παρουσία του εδώ μαζί μας σήμερα. Ε, και για τη διάθεση που έχει πάντα να έρθει εδώ να μας εξηγεί πράγματα. Όταν έφτασα, μιλούσα για ένα θέμα το οποίο επανέρχεται ξανά και ξανά, το, το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων. Είμαι πεπισμένη ότι αν υπάρχει πια σύγκρουση συμφερόντων, αν υπάρχει, είναι μεμονωμένο περιστατικό. Και ούτω ή άλλω οι γνωμοδοτήσει τη ΕΦΣΑ δεν τι φτιάχνει ένα άτομο, τι φτιάχνει ένα πάνελ εμπειρογνωμόνων. Και είναι μια απόφαση που παίρνουν όλοι. Επομένω, ακόμα και αν κάποιο έχει αντιμετωπίζει σύγκρουση συμφερόντων, εγώ ξέρω, γιατί υπήρξα σε τέτοια πάνελ, ε, πάντα υπάρχει κάποιος που έχει τέτοιο θέμα. Οι γνωμοδοτήσει όμω της ΕΦΣΑ δεν είναι η άποψη ενό. Και όταν δεν είναι η άποψη ενό. δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Εμείς έχουμε περιπτώσεις που είναι πάρα πολλά, κάποια θέματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά, όπως η γάμα τάφα όμικρον, οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Και αν δεν πιστεύει η ΕΦΣΑ ότι υπάρχει πρόβλημα με κανένα γάμα ταφόμικρον, δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Ξέρω ότι κάνετε μια έρευνα για το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι αποτελέσματα είχατε, τι απαντήσεις δόθηκαν και τι σκέφτεστε να κάνετε από εδώ και πέρα, ούτως ώστε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια ή δυνατόν. Και αν υπάρχουν υπό, υπόνοιες, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν υπόνοιες, μέχρι εκεί φτάνουμε, υπόνοιες σύγκρουσης συμφερόντων, τι θα γίνει σε αυτήν την περίπτωση. Ξέρω και πιστεύω ότι οι επιστήμονες κάνουν ό,τι μπορούν, προσέχουν πάρα πολύ για να είναι εξάρτητοι. Γιατί είναι θέμα έγκλειστους στην επιστημονική κοινότητα. και εγώ τα λέω αυτά γιατί πιστεύω ότι γενικά δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Εν πάση περιπτώσει, ε, σε αυτή την έρευνα που κάνατε, εσείς τι, σε τι τα καταλήξατε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκοστέτ. Σα ευχαριστώ, Διευθυντή, που ήρθατε ενώπιον της Επιτροπής μας. Η παρέμβασή σα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και συγχαρητήρια για την ποιοτική δουλειά που κάνετε. Για να διευκρινίσετε και να μας φωτίσετε για αποφάσεις που παίρνουμε εμείς και που συχνά είναι πολύ περίπλοκες. Συχνά η δουλειά της, του οργανισμού, του ΕΦΣΑ, ε, δημιουργεί πολεμικές. Μην, μην ξεχνάτε ότι και η επιστήμη δεν είναι αντικείμενο Συνένεση έτσι, απόλυτη συμφωνίας κτλ. Προχωρεί η επιστήμη με κινδύνους, με διαφωνίες. Ε, γι' αυτό συχνά κάνουμε, στήσαμε, στήσαμε και ένα εδόλιο και βάζουμε στο δικαστήριο και στείνουμε, ας πούμε, κατηγορητήριο στην ΕΦΣΑ. Η, η σημασία έχει να υπάρχει διαφάνεια, να υπάρχει επιμερισμός των δεδομένων, ε, να υπάρχει αμεροληψία, γιατί στον επιστημονικό τομέα, όπως και σε άλλους τομείς, σε πολλούς άλλους τομείς, γίνεται πραγματικός πόλεμος ε, ενημέρωσης. Ε, τον βλέπουμε και στα κοινωνικά δίκτυα, πώς λαμβάνει η χώρα. Και όλο αυτό δημιουργεί παραπληροφόρηση, ακόμα και θεωρία συνωμοσία συνέχεια. Αυτές οι μόνιμες αμφισβητήσεις της επιστήμης, στα πλαίσια της δημιουργία δημιουργίας όλο και περισσότερων fake news, είναι επιζήμιο για τη δημόσια συζήτηση και δημιουργεί μια γενικευμένη δυσπιστία στους πολίτες μας απέναντι στην επιστήμη. Και όλα αυτά είναι πολύ λυπηρά, πολύ επιζήμια, γι' αυτό σας υποστηρίζω. Αυτά ήταν σχόλια που έκανα προηγουμένως. Τώρα έχω να κάνω και ένα ερώτημα που δεν αφορά αυτά που είπατε, αλλά είναι ένα θέμα πολύ επίκαιρο και αφορά ε, μία ε, χρωστική ουσία, το ε171, που υπάρχει σε πολλά γλυκά ε, και διερωτώμαστε, είναι επικίνδυνο αυτή η χρωστική. Το Σεπτέμβριο του 2016 η ΕΦΣΑ θεώρησε ότι η χρήση αυτού του, αυτής της χρωστικής δεν είναι επικίνδυνη, αλλά δεν μίλησε για την ε, δυνατή ημερήσια δόση. Όμως στη Γαλλία έχουμε το γαλλικό οργανισμό τροφίμων, ε, ο οποίος ε, μίλησε για επιπτώσεις που δεν είχαν εντοπιστεί πριν και είπε ότι πρέπει να γίνει μελέτη για να χαρακτηρίσουμε το βαθμό επικινδυνότητας που, ε, που συνδέεται με αυτή την ουσία την χρωστική ε171. Ε, διερωτώ με, σκοπεύετε να κάνετε τίποτα για αυτό το θέμα που νομίζω ότι είναι σημαντικό για τον καταναλωτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Μελόρ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ουλρίχ που σήμερα μας χαρίσατε το χρόνο σας ε, και μπορούμε για άλλη μια φορά να συζητήσουμε. Ε, εγώ θα μου επιτρέπετε να ξεκινήσω με μια παρατήρηση. Δηλαδή, ε, νομίζω είστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Το είπατε αυτό και μόνο σας. Εμείς ε, έχουμε προσδοκίες από την ΕΦΣΑ. Η Κομισιόν ε, σας αναθέτει πράγματα. Το Κοινοβούλιο έχει προσδοκίες και ε, περιμένουμε από εσάς ε, ως κράτη-μέλη να τα κάνετε όλα με τους ε, καταπληκτικούς σας επιστήμονες. Εγώ είχα τη δυνατότητα να δω επιτόπου πώς ακριβώς οργανώνεται μια συζήτηση και ένα πάνελ. Μετά δυστυχώς οι πολιτικοί δεν συμφωνούν, σας επιπλήττουν και τι γίνεται πάλι είμαστε εμείς οι οποίοι ψώνουν το δάχτυλο και λέμε μα δεν τα θέλαμε έτσι. Γλυφοσάτη παράδειγμα. Εκεί κατέστη απόλυτα σαφές το τι εννοώ υπήρχαν μελέτες ε, της Μονσάτο, συνοδευτικές, και εγώ σας έστειλα ένα email και σας ρώτησα κατά πόσον ε, αυτές οι μελέτες επηρέασαν το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ που μου απαντήσατε και δείξατε ότι σε όλο αυτό το σωρό και το βουνό των ε, μελετών υπάρχουν δύο-τρεις ε, που είναι πολύ κοντά στη βιομηχανία. Και εσείς ε, μας εξηγήσατε ότι στις περιπτώσεις αυτές είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι προς τα έξω είναι πολύ δύσκολο για σας να πείσετε, να θέσετε σταθερά θεμέλια για την διαφάνεια, για τη συνειδητοποίηση και εδώ θέλω να κάνω την ερώτησή μου. Να ρωτήσω κάτι που αφορά σε αυτό που είπατε κι εσείς. Δηλαδή, η ΕΦΣΑ, ο οργανισμός ΕΦΣΑ, κατ' ουσίαν απαρτίζεται από κράτη-μέλη. Δηλαδή, όλες οι συζητήσεις σε πάνελ εξαρτώνται από την τεχνογνωσία που έχει συγκεντρωθεί στα κράτη-μέλη. Οι συζητήσεις ε, είναι συνάρτηση των μελετών που έχουν καταρτιστεί. Και τελικά πώς γίνεται αυτό. Πώς είναι δυνατόν τα κράτη-μέλη να αισθάνονται περισσότερο ότι είναι δικός μας οργανισμός. Δεν είναι ο απέναντι που αποφασίζει κάτι που δεν θέλουμε καν να το ακούσουμε και που προκαλεί πολιτικές συζητήσεις που απλά είναι κουραστικές. Πώς θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό. Τα κράτη-μέλη να ενστερνιστούν, να αγκαλιάσουν τον ΕΨΑ γιατί με τον τρόπο αυτό μπορούν να υπάρξουν σταθερότερα θεμέλια. Κατόπιν, ρωτήστε, μιλήσατε και για χρήματα και ρωτάω για πόσα, για πόσα συζητάμε, ποια είναι τα κονδύλια που χρειάζεστε επιπρόσθετα έτσι ώστε να μπορέσετε να τεκμηριώσετε καλύτερα την επιστημονική σας εργασία. Και ίσως και πέρα από τη χρηματοδότηση να υπάρχουν και άλλες δυνατότητες για το πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε εμείς ως βουλευτές. Και αν μπορέσουμε αυτό να το κάνουμε με τα κράτη-μέλη από κοινού, αυτό θα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Ρόιταμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που ήρθατε που προσπαθείτε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις μας. Καταρχάς να κάνω μια δήλωση. Ελπίζω όλοι να συμφωνήσετε εδώ στην Επιτροπή μου αυτή. Είναι πολύ σημαντικό να βασίζουμε τις αποφάσεις μας, ειδικά σε αυτήν την Επιτροπή, στην επιστήμη. Και με μεγάλη χαρά είδα, πριν από καμιά δύο εβδομάδες, την πορεία της επιστήμης στον υπόλοιπο κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό και τις πολιτικές αποφάσεις να τις βασίζουμε περισσότερο στην επιστήμη και να μην λαμβάνονται με δημαγωγικό τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό και εδώ. Χαίρομαι λοιπόν που έχουμε αυτό το φορέα την ΕΦΣΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπατε και στην ε, εισαγωγική σας παρέμβαση, είναι πολύ σημαντικό να ακούμε τις κριτικές, να κάνουμε καλύτερες διαδικασίες, να είμαστε πιο διαφανείς, ε, να κάνουμε έλεγχο του σύγκρου ε, συμφερόντων ποιοτικέ έρευνε και επαρκή χρηματοδότηση κυρίω. Είναι κάτι που συχνά παραβλέπουμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό για την ΕΦΣΑ. Έχω την αίσθηση μερικέ φορέ ότι κάποια από τα αποτελέσματα, κάποια από τα συμπεράσματα της ΕΦΣΑ ή τα πορίσματα της ΕΦΣΑ δεν τα συμμερίζονται όλοι οι πολιτικοί. Οκ, γίνεται. Όμω, η αντίδραση ε, κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων ή της αμφισβήτησης, μάλλον η ε, της αμφισβήτησης ΕΦΣΑ είναι πολύ επικίνδυνο. Μπορεί να διαφωνείτε με τα γάματα φόμικρον, αλλά το να αμφισβητείτε την ΕΦΣΑ είναι πολύ επικίνδυνο τελικά. Και να χρησιμοποιεί το επιχείρημα της ε, διαφάνειας ε, και της σύγκρουσης των συμφερόντων για να κατηγορήσει την ΕΦΣΑ είναι κακό. Θα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι αντίθετα και να αισθανόμαστε τυχεροί που έχουμε ένα επιστημονικό φορέα ο οποίος δεν χρειάζεται να κάνει πολιτική συζήτηση για επιστημονικά θέματα. Κάτι που είναι πολύ επικίνδυνο. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι αυτό που έχουμε είναι πολύτιμο. Τώρα μια πιο συγκεκριμένη ερώτηση για τα έγγραφα της Μονσάντο. Για την γλυφοσάτη που έχει μελετηθεί πάρα πολύ. Ε, είναι από τα πιο μελετη... Ε, Είναι ένα από τα ζυζανιοκτώνα οποία... για τα οποία υπάρχουν πάρα πολλά έγγραφα. Ε, τώρα ε, μάθαμε ότι κάποιες από τις μελέτες της επηρέασε η Μονσάντο. Θα αναθεωρήσει τις, τα πορίσματά της η ΕΦΣΑ μετά από αυτές τις αποκαλύψεις για την γλυφοσάτη. Και τι θα, τι θα διδαχθεί για το μέλλον. Και ποιες είναι οι συνέπειες για το εγγύς μέλλον από αυτές τις αποκαλύψεις. Η κυρία Γκέρλιν. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον, ε, Διευθυντή της ΕΦΣΑ που ήρθε. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση και τον τρόπο που παρουσιάσατε τα θέματα. Είναι πραγματικά αναζωογονητικό ε, να έρχεται κάποιο εδώ και να μπει στο ψητό κατευθείαν παρά να το πάει γύρω-γύρω, ας πούμε. Οι περισσότερες ήταν καλές ερωτήσεις ε, και απαντήσατε σωστά και ε, στα, πάνω στα θέματα που θέσατε. Με βάση αυτά που ακούσαμε χθε από τον Επίτροπο Άνδριου Κάιτης, όπου ξεκαθάρισε ότι θα εξετάσει ε, το θέμα της αναθεώρησης του General Food Law, προτεραιότητά του. Και η ΕΦΣΑ δημιουργήθηκε από αυτό το νομοσχέδιο για το, γενικό νομοθέτημα για τα τρόφιμα, το General Food Law. Ε, και μια και θα υπάρξει αναθεώρηση και καθώς θα προχωράει θα πρέπει να αναθεωρηθεί άρδιν η ΕΦΣΑ. Ίσως θα είναι μια ευκαιρία λοιπόν και για σας και για μας για να αναλύσουμε κριτικά ε, σε ποιο βαθμό η ΕΦΣΑ κάνει τη δουλειά που θέλουμε να κάνουμε. Που θέλουμε να κάνει. Εγώ παρεμπιπτόντως να σας πω ότι κάνει θαυμάσια δουλειά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβληματικά σημεία και ότι δεν θα ήθελα να ασκήσω κριτική σε κάποια θέματα. Έχετε 10 επιστημονικά πάνελ καταρχάς ε, αυτή τη στιγμή. Ε, και η Επιστημονική Επιτροπή αποτελείται από τους προέδρους των πάνελ. μερικές φορές τα μηνύματα για τις επιστημονικές αποφάσεις φιλτράρονται από αυτά τα πάνελ ε, και εγώ συναντήθηκα μάλιστα με κάποιους οι οποίοι ήταν σε πάνελ της ΕΦΣΑ στο παρελθόν που τους αποθαρρύνει το γεγονός. Γιατί το γεγονός ότι τους ασκούν διάφοροι κριτικές, ας πούμε, ε, το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή μας κτλ. για τη δουλειά που κάνανε. Είναι δύσκολο να πει ένα επιστήμονα 55 ας πούμε, ο οποίο δεν δούλεψε ποτέ για τη βιομηχανία. Εγώ συναντήθηκα με κάποιον ε, τι προάλλε που του ασκήσαν κριτική γιατί ένα τμήμα του διδακτορικού του που το έχει κάνει πριν 30 χρόνια χρησιμοποίησε δεδομένα από μια μεγάλη χημική εταιρεία. Αυτό ήταν άδικο γιατί στην πραγματικότητα ποτέ δεν δούλεψε για αυτή τη χημική εταιρεία, απλώ χρησιμοποίησε δεδομένα. Επομένως, ε, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε για αναθεωρήσεις. Τώρα, ποια είναι η ερώτησή μου συγκεκριμένα. Αυτό, αυτή η νομοθεσία για τα τρόφιμα, αυτή η αναθεώρηση της νομοθεσίας, πού βλέπετε να πηγαίνει. Έχει, θα παίξει κάποιο σημαντικό ρόλο σε αυτή την αναθεώρηση η ΕΦΣΑ. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε την ευκαιρία για να αντιμετωπίσετε κάποια από τα θέματα που εντοπίσατε και εσείς στην παρέμβασή σας. Και το θέμα της χρηματοδότησης επίσης, γιατί αν θέλουμε περισσότερα πράγματα να κάνει η ΕΦΣΑ, ίσως θα πρέπει να αλλάξουμε το μοντέλο χρηματοδότησης. Παραδείγματο χάρη, ας πούμε, να καταβάλλονται τέλη για κάποια πράγματα, για κάποιες δουλειές που κάνει η ΕΦΣΑ. Ευχαριστώ. Κύριος ε, Χάουσλινγκ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ε, είχαμε στην Επιτροπή Γεωργίας μια πολύ ζωντανή συζήτηση και κατ' ουσίαν εκεί συζητήσαμε το ίδιο θέμα που αυτό που αναφέρετε κι εσείς. Ε, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη έναντι της εμπιστοσύνης και κάποτε αυτό πρέπει να γίνει αποδεκτό. Και εδώ ξεκινάει η κριτική μου. Η ανεξάρτητη επιστήμη η οποία υπηρετεί, προσφέρει κάτι, αυτό δεν υπάρχει πια, τέλος. Και βέβαια δεν φταίτε εσείς γι' αυτό. Ε, φταίει το ότι τα πανεπιστήμια όλο και περισσότερο εξαρτώνται από χρηματοδότηση από τρίτους ε, φορείς. Ε, άρα δηλαδή αυτοί οι ανεξάρτητοι επιστήμονες δεν υπάρχουν αυτοί. Αυτό το ρόλο θα έπρεπε να τον αναλάβει ο ΕΦΣΑ και με τους ε, ανεξάρτητους επιστήμονες να προβαίνει σε πιο ουσιαστική έρευνα. Ε, τώρα εσείς με τα μέσα που διαθέτετε το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι κατά πόσον αυτά που ε, θεσπίζονται συμβατίζουν με την επιστήμη. Αλλά αμυγός ανεξάρτητες επιστημονικές μελέτες αυτές δεν μπορείτε να τις εκπονήσετε. Νομίζω το είπε και ο σε συνάδελφός μου. Εγώ πιστεύω ότι πολλοί θα σας διέθεταν τα κονδύλια τους ευχαρίστω αν πραγματικά ήταν σίγουροι ότι είσαστε ανεξάρτητοι. Γνωρίζετε τη συζήτηση που γίνεται στις Ηνωμένε για τη γλυφοσάτη. Ε, γνωρίζετε κατέστη σαφές ότι η Μονσάντο επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το τι γράφεται, το τι δημοσιεύεται και επίσης ότι η Μονσάντο έχει και άμεση επαφή ε, και με εκείνους που είναι αρμόδιοι για την αδειοδότηση. Άρα φαντάζομαι όλοι συμφωνείτε ότι δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιστημονική μελέτη σε σχέση με τη γλυφοσάτη. Να ρωτήσω και κάποια άλλα πράγματα που δεν τα δείξατε. Πρώτον, τα νέο νοικοτονοειδή γνωρίζετε ότι αυτά τα νεονικοτονοειδή ε, είναι ιδιαίτερα ε, επίμαχο σε σχέση με τη μελισσοκοπία και θέλω να ρωτήσω, εσείς πότε υπολογίζετε να αποσυρθούν οι επικίνδυνες ουσίες και θα τα τεκμηριώσετε αυτά επιστημονικά. Κατόπιν, νέες μέθοδοι καλλιέργειας και εκτροφής. Η ΕΦΣΑ τοποθετήθηκε πρόσφατα, θα εξηγήσετε λιγάκι και τους κινδύνους, γιατί αυτό που με εκνευρίζει είναι ότι μέχρι τώρα δεν έχει τοποθετηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι επικίνδυνες τεχνολογίες ε, πώς ακριβώς ε, συντάσσονται, ποιες είναι. Τέλος, ε, σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, αυτά που λέγονται όλα με θλίβουν. Και θέλω να σας πω, εσείς ε, θα τοποθετηθείτε επ' αυτού με σαφήνεια, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πραγματικά υστερεί στο θέμα αυτό σε σχέση με άλλους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καπούτο. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε και ευχαριστώ τον Διευθυντή της ΕΦΣΑ για τη διάθεσή του να συζητήσουμε. Θα ήθελα να κάνω ένα ειδικό, ιδιαίτερο ερώτημα. Πριν από λίγο, μια έκθεση της ΕΦΣΑ επιβεβαίωσε ότι φτάνει στην Ευρώπη μια νέα ασθένεια των βοηδών την ο, μεταδοτική οζόδη ε, δερματίτιδα που ξεκίνησε από την Αφρική, ε, πέρασε στην ε, Τουρκία, στα Βαλκάνια και έφτασε έως την Ρωσία. Ε, είναι μεταδοτική αρρώστια στα, στα βοηδή που μεταδίδεται από τα έντομα. πρέπει να υπάρχει αυστηρότος έλεγχος από τις υγειονομικές αρχές και να υπάρχει και σωστή εκστρατεία εμβολιασμού. Μόνο αυτό είναι ε, αποτελεσματικό. Μιλάμε για έναν ιό POX που μπορεί να ζήσει ε, για ένα αρκετό διάστημα μέσα στην, ε, στον οργανισμό του ζώου. Πώς εκδηλώνεται η αρρώστια. Έχουμε όζους στο δέρμα και έχουμε ε, θνησιμότητα από 5 45%. Έχουμε τεράστιες οικονομικές απώλειες για τους ακτινοτρόφους και σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των ζώων. Είναι κατεπήγον λοιπόν να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για την νέα αυτή αρρώστια, ειδικά σε ό,τι αφορά το κίνδυνο και την, τα προβλήματα που θέτει στην, διατροφική ασφάλεια, ε, τα παράγωγα προϊόντα από το βόλιο κρέας και τις πιθανές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Ευχαριστώ. Κυρία Γκούτελαντ, ποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο? Κυρία Γκούτλαντ, σας ευχαριστώ για αυτή τη δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων και για την εισήγησή σας. Με ενδιαφέρει ένα θέμα που έφυξαν και άλλα μέλη, τα νεονικοτινοειδή και αυτό γιατί από τους μελισσοκόμους ακούω πολλά για προβλήματα με τις μέλισσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μέσα σε λίγα χρόνια ε, έχουμε υψηλή θνησιμότητα μελισσών και σίγουρα τα παρασιτοκτόνα και τα νεονικοτινοειδή είναι ένας παράγοντας. Στη Σουηδία η αρχές διαπίστωσαν ότι υπάρχει, υπάρχουν επιπτώσεις και στις άγριες μέλισσες. Σε αυτό το συμπέρασμα φτάσαμε. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε ποια είναι τα δικά σας συμπεράσματα για τα νεονικοτινοειδή, γιατί είναι κάτι το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί προτεραιότητα. Ο κύριος Ντεμέρσμακερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί σήμερα μπορούμε να προδούμε σε μία ανταλλαγή απόψεων. Εγώ είμαι υπέρμαχος των θέσεων της ΕΦΣΑ και της ίδιας της ύπαρξής της και θεωρώ ότι πρέπει να διαθέτουμε έναν τέτοιο οργανισμό και εγκρίνω και τις μεθόδους της πέρσι βρέθηκα στην Πάρμα και ε, πολλά ζητήματα κατέστησαν απόλυτα σαφή για μένα. Υπάρχει ανάγκη διασφάλισης διαφάνειας και ανεξαρτησίας για να κρατήσετε την εμπιστοσύνη της κοινή γνώμης και για να απομακρύνετε και τη δυσπιστία της κοινή γνώμης σε σχέση με τους κινδύνους για την υγεία. Αν μιλάμε για κινδύνους για την υγεία ή καρκινογόνες ουσίες, εσείς θα πρέπει να έχετε ακόμα μεγαλύτερη διαφάνεια, αλλά υπάρχουν ορισμένα όρια και μας είπατε πού βρίσκονται αυτά τα όρια. Νομίζω ότι τουλάχιστον θα πρέπει να καταστήσετε σαφές προς τον έξω κόσμο Ποια ήταν η συνεισφορά της Μονσάντο ε, κατά την τελική γνωμοδότηση για τη γλυφοσάτη. Νομίζω ότι αυτές τις πληροφορίες θα πρέπει να τις κοινοποιήσετε. Και έχω και δύο ερωτήματα στις εισαγωγικές παρατηρήσεις μας ε, Μιλήσατε για την υποστήριξη της ΕΦΣΑ προς τους επιστήμονες έτσι ώστε να προβούν σε μια νέα αξιολόγηση. Σταθήκατε σε αυτό κατά την εισήγησή σας, αλλά μπορείτε να μας μιλήσετε για τα υπέρ και τα κατά αυτού του προτύπου υποστήριξης που εφαρμόζεται στην, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Ο κύριος Τέρζη από την Επιτροπή, αν έχει κάτι να προσθέσει. Όχι, εντάξει, αν δεν έχετε λόγο να λάβετε το, το λόγο. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ούρλ για να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις, πολύ τροφή για σκέψη. Θα είναι δύσκολο να είμαι σύντομος. Θα με σταματήσετε αν χρειαστεί. Ε, καταρχήν να ευχαριστήσω την κυρία Αγιούζο για τη συνεχή υποστήριξη, γιατί είσαστε και ο σύνδεσμός μας. Μιλήσατε για ε, σύγκρουση συμφερόντων. Αυτό που προσπαθούμε είναι να έχουμε μία δημόσια διαβούλευση για τη νέα πολιτική ανεξαρτησίας που θα συζητήσουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο τον Ιούνιο. Υπάρχει ανοιχτή διαβούλευση, γι' αυτό θα θέλαμε και εσείς να συνεισφέρετε στην πολιτική μας γιατί ασχοληθήκαμε και με ζητήματα που προέρχονται από το Κοινοβούλιο. Ότι πώς ορίζουμε δηλαδή τα συμφέροντα έτσι ώστε να μην είναι συγκρουόμενα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης συνέταξε ένα έγγραφο για την πολιτική ανεξαρτησίας από το 2011 και η έκβαση αυτής της μελέτης ε, είναι, έχει δημοσιοποιηθεί. Η πολιτική είναι αποτελεσματική, δηλαδή προστατεύει από σύγκρουση συμφερόντων. Είναι μεγάλος ο γραφειοκρατικός πόρτος γιατί ε, έχουμε μία ετήσια αποτίμηση 700 ε, δηλώσεων συμφερόντων. Βλέπουμε ποια είναι τα συμφέροντα Έχουμε νέα κατηγορίες από χρηματοοικονομικές μέχρι την απασχόληση, έρευνα, πνευματικά δικαιώματα και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα βρίσκεται στις δηλώσεις συμφερόντων και είμαστε πεπισμένοι ότι έχουμε οικοδομήσει ένα εύρωστο σύστημα, ίσως το πλέον εύρωστο, στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αλλά μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω. Γι' αυτό υπάρχει η διαδικασία της δημόσιας ε, διαβούλευσης, έτσι ώστε το καλοκαίρι ίσως να καταρτήσουμε μια νέα πολιτική. Κυρία Γκροστέτ, για το E171, διοξίδιο του τιτανίου, θα γνωμοδοτήσουμε. Και υπάρχει το θέμα της συμπίκνωσης, δηλαδή το νανοκλάσμα αυτό, το νανοσωματίδιο που χρησιμοποιείται ε, στο διοξίδιο του τιτανίου και η ένας ευρωπαϊκός οργανισμός, εκπώνησε μία μελέτη για το κατά πόσο υπάρχουν τοξικολογικά ευρήματα έτσι ώστε να γίνει μια νέα αποτίμηση του, ε, διοξιδίου του Τιτανίου. Ήρθαμε σε επαφή με τον ε, γαλλικό οργανισμό. Είδαμε αυτή τη μελέτη για να δούμε κατά πόσο θα πρέπει να αλλάξουμε την περιεκτικότητα σε διοξίδιο του Τιτανίου τα στοιχεία δεν είναι πιστικά, χρειαζόμαστε επιπρόσθετα στοιχεία για να έχουμε περισσότερες γνώσεις για αυτό το νανοκλάσμα του διοξιδίου του τιτανίου. Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο της ΕΦΣΑ και της ΑΝΣΕΣ, μιας πολύ μεγάλης ε, επιστημονικής κοινότητας της Ευρώπης και νομίζω τα καταφέραμε πολύ καλά με αυτή τη συνεργασία Άνσες και Εύσα. Δεν θα μιλήσω γερμανικά. Για στο ερώτημά σας πώς η ΕΦΣΑ μπορεί να γίνει δική μας ΕΦΣΑ πώς μπορεί να υπάρχει ένα μεγαλύτερο ιδιοκτησιακό καθεστώς, ένας προσετερισμός δηλαδή, έχει μεγάλη σημασία γιατί η ΕΦΣΑ έχει ένα διαφορετικό διοικητικό συμβούλιο. Δεν υπάρχουν τα κράτη-μέλη στο διοικητικό συμβούλιο. Η ΕΦΣΑ έχει 14 εκπροσώπους, είναι έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μετά την ε, σπογγόδη εγκεφαλοπάθεια των βοηδών, καταρτίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει ένα ευρύ φάσμα κάλυψης των ασθενειών. Εμείς προωθούμε την επιστημονική συνεργασία όλα τα κράτη βρίσκονται στο συμβουλευτικό φόρουμ, τέσσερις φορές το χρόνο συνερχόμαστε και δημιουργούμε την Ευρωπαϊκή Ατζέντα Αξιολόγησης Κινδύνου, όπου εντάσσουμε project ε, όπως ε, ζήτησε και ο Γερμανικός Οργανισμός για ε, μια διαδικασία ιχνηλάτησης ή του Βρετανικού Οργανισμού για τα ιογενή στοιχεία και πληθώρα άλλων οργανισμών. Το Κοινοβούλιο μπορεί να μας υποστηρίξει στις εκλογικές σας περιφέρειες δηλαδή, γιατί χρειαζόμαστε μια πολιτική υποστήριξη από τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε και σε δυσμενείς οικονομικούς καιρούς οι οργανώσεις των κρατών μελών να επιτρέπουν στους ανθρώπους να εργάζονται για αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Είναι πολιτικό ε, ε, το ζήτημα και ακούμε από τις οργανώσεις των κρατών μελών που θέλουν ε, να συνεργαστούν με την ΕΦΣΑ, αλλά υπάρχουν περικοπές κατά 20-30% και χρειάζονται την επιστημονική τους κοινότητα στην πατρίδα τους. Εάν αυτό συνεχιστεί, δεν θα υπάρχει πια βιώσιμο ε, πρότυπο της ΕΦΣΑ. Μπορούμε να κλείσουμε τον οργανισμό αυτό. Γι' αυτό χρειαζόμαστε πολιτική υποστήριξη. Είναι ένα θέμα που αφορά την Ευρώπη καθαρά την Ευρώπη. Και γνωρίζουμε ότι αυτή η συζήτηση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Ως προς το χρηματικό, δεν έχουμε ε, υπολογίσει μέχρι το τελευταίο ευρώ είναι οι ανάγκες, αλλά πρόκειται για 20 εκατομμύρια ευρώ που πρέπει να καταβληθούν στα κράτη-μέλη. Και πώς αυτό διαφέρει από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων η αίμα έχουμε να κάνουμε με ε, ένα μέγεθος δύο φορές της ΕΦΣΑ, αλλά ε, προπολισμό τέσσερις φορές της ΕΦΣΑ. Καταβάλουν λοιπόν τα χρήματα για τη συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, την αίμα 140 εκατομμύρια ευρώ που διανέμει αίμα στα κράτη-μέλη, το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς. Άρα πολιτικά θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε την ΕΦΣΑ, να υπάρχουν τέλη, ειδικά τέλη ή οτιδήποτε άλλο και για τη βιωσιμότητα αυτού του προτύπου και για να έχουμε πρόσβαση στις, στην καλύτερη τεχνογνωσία της Ευρώπης. Μιλήσατε και για τα έγγραφα της Μονσάντο και την επιρροή τους στην ε, αξιολόγηση της γλυφοσάτης. Από όσο γνωρίζουμε, ε, μιλάμε για δύο έγγραφα όπου η εσωτερική αλληλογραφία δείχνει ότι ίσως η Μονσάντο είχε, Μονσάντο είχε συμφέροντα για κάτι τέτοιο, αλλά αναφέρεται και η σχέση των συγγραφέων με την Μονσάντο. Δεν υπάρχει ένα στοιχείο έκπληξης και είναι δύο οι μελέτες από τις 700. Άρα πρόκειται για ένα περιορισμένο στοιχείο, δύο μελέτες από τις 700. Δεν είχαμε πρωτογενή στοιχεία, δηλαδή οι επιστήμονες αναθεώρησαν τα στοιχεία άλλων επιστημόνων, που είναι μια τρέχουσα πρακτική εμείς. Ως αξιολογητές κοιτάμε την πρώτη ύλη γιατί θέλουμε να φτάσουμε στα δικά μας συμπεράσματα. Άρα εμείς ε, λαμβάνουμε τα πρωτογενή στοιχεία και τα επεξεργαζόμαστε. Δεν θεωρούμε ότι κάτι θα αλλάξει στην ε, αξιολόγηση της γλυφοσάτης δεν υπάρχει λόγος ε, έλλειψης εμπιστοσύνης. Ίσως υπάρξουν νέες εξελίξεις, όμως ως ΕΦΣΑ είμαστε οι θεματοφύλακες ε, της επιστήμης. Αν σπηλωθεί η επιστήμη, τότε μπορούμε να την ξεχάσουμε. Χρειαζόμαστε αμερόληπτα επιστημονικά στοιχεία. Ε, κύριε Χάισλινγκ, είπατε ότι εγώ θεωρώ ότι η επιστήμη είναι η μόνη απάντηση, είναι μια παγκόσμια αλήθεια. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε έναν οργανωμένο σκεπτικισμό. Μπορεί να μεταλλαχθεί αύριο, αλλά αυτή είναι και η δύναμη της επιστήμης που μπορεί να ε, παραποιηθεί ε, εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε δογματισμούς και ιδεολογίες. Θα πρέπει να υπάρχει επεξεργασία στοιχείων για να αποτιμήσουμε τα φαινόμενα της φύσης και της κοινωνίας. Είναι το καλύτερο μέσο που διαθέτουμε. Γιατί η εναλλακτική θα ήταν η μεσαιωνική σκέψη. Δεν υπάρχει εναλλακτική, γι' αυτό η διαδικασία αυτή θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα εύρωστη. Μπορούμε να επικρίνουμε την επιστήμη. Μιλήσατε για την εμπορικοποίηση των πανεπιστημίων. Ποιος χρηματοδοτεί τα πανεπιστήμια. Ο ειδικό τομέα. Αλλά αυτό είναι ένα πολιτικό ερώτημα. Ε, πώς διαχειρίζεστε την επιστήμη. Είναι ένα θέμα πολιτικών διαπραγματεύσεων. Επίσης, θέσατε και το ερώτημα του τι μαθαίνουμε. Θα πρέπει να επαγρυπνούμε περισσότερο ως προς τις πηγές μας, τις πρωτογενείς πληροφορίες και την ανάλυση των στοιχείων. Όταν έχουμε αποδεικτικά στοιχεία και εμείς έχουμε το σχέδιο Προμηθέας που ασχολείται με τη συλλογή και επεξεργασία αποδεικτικών στοιχείων που είναι διαφανή και αναπαράξιμα και τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Κυρία Γκέρλινγκ, μιλήσατε για το, το εγχείρημα Refit, το οποίο διέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς συμμετέχουμε στη διαδικασία Refit. Η εντολή λυγεί φέτος και για μας αυτό αποτελεί ευκαιρία να θίξουμε ζητήματα για την ε, βιωσιμότητα, τη σύσταση της επιστημονικής κοινότητας, τη διάρκεια των πάνελ για τρία χρόνια, ίσως περισσότερο, για να μειώσουμε και το διοικητικό φόρτο. Άρα θα δώσουμε και τα δικά μας στοιχεία και κάθε έξι χρόνια η ΕΦΣΑ υπόκειται σε εξωτερικό έλεγχο διανόμου. Το 2012 έγινε η τελευταία εξωτερική αξιολόγηση, άρα το 2018 ε, θα έχουμε την επόμενη και αποτιμούμε τον αντίκτυπο της ΕΦΣΑ στην ε, διατροφική, στην, ε, ως προς την υγεία των τροφίμων και αποτιμούμε κατά πόσο είναι το καλύτερο πρότυπο τουλάχιστον μέχρι το 2020, ίσως μέχρι μέσα σε 15 χρόνια να βρούμε ένα νέο τρόπο αποτίμησης των κινδύνων στην Ευρώπη. Η ε, κύριε Χόισλινγκ, ε, μίλησα για την επιστήμη και το ρόλο της επιστήμης καθώς και την ευαλωτότητα της επιστήμης. Και αυτό που έχει σημασία είναι κατά πόσο παραποιούνται τα στοιχεία. Ως προς τη Μονσάντο πιστεύω ότι σας απάντησα. Ναι, μας απασχολεί το ζήτημα φυσικά. Θέλουμε να επαγρυπνούμε ως προς τα νεονικοτινοειδή. Είχαμε μία επιστημονική μελέτη το 2012 και το 2013 και είχαμε και συνενετικά στοιχεία τα οποία δημοσιοποιήθηκαν το 2016. Και τώρα γίνεται μία επανεκτίμηση των ε, νέων, για τα νέα νέων νοικοτινοειδή και τα στοιχεία θα δημοσιευτούν τον Νοέμβριο 2017. Δεν θα αποφασίσει η ΕΦΣΑ κατά πόσο αυτές οι ουσίες επιτρέπονται ή όχι. Η Επιτροπή θα το κάνει αυτό και τα κράτη-μέλη, αλλά θα τους υποστηρίξουμε με τα νέα επιστημονικά στοιχεία σε σχέση με τους κινδύνους νεονικοτινοειδών. Ως προς τη νέα διαδικασία καλλιέργειας, είχαμε ένα ε, έγγραφο ε, το οποίο ε, δημοσιοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προηγούμενη Παρασκευή και βλέπουμε το θέμα κατά περίπτωση και βλέπουμε κατά πόσο αυτή η αποτίμηση κινδύνων θα πρέπει να υπόκειται στον ε, κανονισμό για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Αυτό θα το δουν οι νομοθέτες, όχι οι ε, επιστήμονες. Σε σχέση με τους ε, ενδοκρινικούς διαταράκτες, ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει κριτήρια και η ΕΕΦΣΑ προβάλλει ένα έγγραφο κατευθυντηρίων γραμμών μαζί με την ΕΚΑ να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία για τα παρασιτοκτόνα και τα φυτοκτόνα. Προς τον κύριο Καπούτο, ναι, υπάρχει αυτό το θέμα της οζόδους δερματίτιδας στη Νότια Ευρώπη, στην Ελλάδα, στις Βαλκανικές χώρες, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος και στην Κροατία και γίνεται εμβολιασμός και γι' αυτό δεν διαδόθηκε η ασθένεια και ελέγχουμε και δίνουμε στην Επιτροπή στοιχεία για να δούμε πόσο, κατά πόσο μπορούμε να αναχαιτήσουμε αυτή την ασθένεια, αλλά προβαίνουμε σε διαχείριση κινδύνου που γίνεται από τα κράτη-μέλη και την Κομισιόν. Well, on, on bee health Ως προς τα δεν ξέρω κατά πόσο απάντησα. Νομίζω ότι δεν ξέχασα κανέναν. Πώς η ΕΦΣΑ υποστηρίζει άλλους επιστήμονες. Αυτό προσπαθούμε να δούμε είναι η επιστήμη να είναι διαφανή σε σχέση με στοιχεία και μεθοδολογίες ώστε να μπορέσει να έρθει οποιοδήποτε να ε, κατεβάσει τα στοιχεία από τον ιστότοπό μας και να δει και να προβεί σε μια νέα αξιολόγηση αν θέλει. Θέλουμε να είναι αναπαράξιμη η αξιολόγηση κινδύνου. Είναι φιλόδοξος ο στόχος, δεν θα γίνει αύριο το πρωί. Χρειάζεται συνεργασία από τη βιομηχανία, από τα σωστά μέσα είναι μέρος της στρατηγικής ΕΦΣΑ 2020, ε, αλλά θα φτάσουμε σε αυτό το στόχο για να είναι αναπαράξιμη η αξιολόγηση κινδύνου. Και χαιρόμαστε γιατί υπάρχει αυτή η αξιολόγηση και ο φιλόδοξος στόχος. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ε, για την ανταλλαγή απόψεων. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ήταν ε, αυτή η ανταλλαγή. Ε, και έτσι λοιπόν περνάμε στο επόμενο θέμα, αγαπητοί συνάδελφοι, το οποίο επόμενο θέμα είναι τα φυτικά έλαια. Και έχουμε βεβαίως και την ΕΦΣΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα φυτικά έλαια. ξεκινάμε με την ΕΦΣΑ. Λοιπόν, θα ακούσουμε πρώτα την τοποθέτηση της ΕΦΣΑ. Λοιπόν, είμαστε όλο αυτιά. Έχετε το λόγο. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα να έρθουμε σήμερα εδώ για να σας εξηγήσουμε την αξιολόγηση κινδύνου για τα φυτικά έλα και για τους ε, επιμολυντές. 16 Μαΐου δημοσιεύσαμε την επιστημονική μελέτη ε, σχετικά ε, με τους κινδύνους που μπορεί να υπάρχουν στο ραφιναρισμένο έλαιο. Τους επιμολυτές, ε, τους αξιολογήσαμε, το MCPD, τα αποκαλούμε 3 και 2 MCPD και εξετάσαμε επίσης ε, και τους ε, εστέρες λιπαρών εξαίων. Διαπιστώθηκε ότι οι επιμολυντές 3 και κυρίως 2 MCPD προκαλούνται κατά την βιομηχανική παραγωγή των υδρο, των υδρολιμένων φυτικών πρωτεϊνών. Όσον αφορά λοιπόν ε, αυτές τις ε, δύο ουσίες, αυτές ε, ορίζονται τα ανώτατα όρια τους στον κανονισμό του 2006 και αργότερα διαπιστώθηκε ότι αυτοί οι δύο επιμολυντές συν οι στέρες του γλυκιδόλης παρουσιάζονται στα λιπαρά έλαια. Ο στόχο είναι όμως ότι, μάλλον υπάρχει το εξή ότι προτίστε ουσίε για να γίνονται αυτές οι ουσίε πιο βρώσιμες. Ε, υπάρχουν πολλά στοιχεία που συγκεντρώσαμε σε πειράματα σε ζώα αλλά και από την βιβλιογραφία. Επίσης ε, αξιολογήσαμε την έκθεση των επιμολυντών και λάβαμε υπόψη μας ε, την κατάσταση που επικρατεί στα κράτη-μέλη, στη βιομηχανία. Λάβαμε υπόψη μας και τα δεδομένα που υπήρχαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τα στοιχεία κατανάλωση που υπέβαλαν τα κράτη-μέλη. Για να μπορέσουμε λοιπόν να εξηγήσουμε την διατροφική έκθεση εξετάσαμε διάφορες ομάδες, παιδιά μέχρι ενός έτους, έφηβους και ενήλικες. Και κατόπιν υπολογίσαμε ή φτιάξαμε ένα θεωρητικό σενάριο όπου ε, χρησιμοποίησαμε μια συγκεκριμένη φόρμουλα. Με βάση λοιπόν την αξιολόγηση κινδύνου, τα υψηλότερα επίπεδα αυτών των επιμολυντών διαπιστώθηκαν στα φυτικά έλαια και στα λίπη. 6 μέχρι 10 φορές ε, υψηλότερο το επίπεδο σε φινικέλαιο και σε ε, λιπαρά, σε λείπει φινικελαίου. Βέβαια υπάρχει ε, μεγάλη διακύμανση στις ομάδες ε, για τα μικρά παιδιά. Ε, η μεγαλύτερη έκθεση είναι στα φυτικά έλα, στους έφηβους και στα, στους ηλικιωμένους. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει τόσο κίνδυνος κυρίως και στη μαργαρίνη και σε άλλα προϊόντα. Στην τελευταία κατηγορία επικίνδυνη ουσία στη μαργαρίνη, στις βάφλες, σε προϊόντα πατάτας και επίσης και σε επικαλύψεις της ε, σοκολάτας. Αυτά λοιπόν όλα διαπιστώθηκε ότι ε, μπορούν να είναι επικίνδυνα για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Και με βάση μελέτες σε ζώα αξιολογήσαμε ότι η έκθεση το 3-MCPD καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής αυτό μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στον οργανισμό. Ε, η καθημερινή ε, ανεκτή μερίσια λήψη κατά 0,8 ανάλογα με το βάρος. Ε, αυτό καθορίστηκε για την 3, ε, τον επιμολυντή 3MCPD. Κατόπιν για τους εστέρες διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι οι εστέρες γλυκιδόλης είναι καρκινογόνες ουσίες. Για άλλες ε, καρκινογόνες ουσίες αυτές θα μπορούσαν να προσβάλλουν το DNA και να προκαλέσουν καρκίνο και διαπιστώσαμε ότι οι εστέρες γλυκιδόλης μπορούν να προκαλέσουν μεγαλύτερη εμφάνιση καρκινογόνων όγκων. Θελήσαμε λοιπόν να ορίσουμε και να καθορίσουμε το περιθώριο της έκθεσης. Για αυτές τις ενώσεις, τους εστέρες γλυκυντόλης, το περιθώριο ε, προκαλεί πράγματι ανησυχία για όλους τους νέους ε, με μεσοσταθμική έκθεση και για καταναλωτές με υψηλότερη έκθεση σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Κυρίως η έκθεση σε εστέρες για μωρά είναι 10 φορές ε, μεγαλύτερη, ε, κυρίως όταν τα παιδιά καταναλώνουν παιδικό γάλα. Για τον επιμολυντή 2MCPD δεν μπορέσαμε και να καταλήξουμε γιατί δεν έχουμε απαραίτητα δεδομένα. Για τον επιμολυντή 3MCPD η έκθεση η έκθεση ξεπερνάει την ε, ανοιχτή ημερήσια λήψη κυρίως στην περίπτωση των παιδιών που λαμβάνουν μόνο παιδικό γάλα. Ε, έξι μήνες αργότερα, Τζέκφα, που είναι η κοινή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για πρόσθετες ουσίες στα τρόφιμα αξιολόγησε τους εστέρες του 3-MCPD και τους εστέρες γλυκιδόλης και δημοσίευσε τα αποτελέσματα. Ο οργανισμός αυτός και η ΕΚΦΑ συμφώνησαν σε μία μελέτη που έλαβε υπόψη της ε, την αξιολόγηση αλλά και τις αρνητικές επιπτώσεις των επιμολυντών. Μετά από αυτή τη μελέτη και λαμβάνοντας υπόψη νέες εξελίξεις της μεθόδου. τώρα πλέον εργαζόμετα για τον επιμολυντή 3MCPD και την εργασία μας θα τη δημοσιάσουμε στο τέλος του έτους. Για τους εστέρες γλυκυδόλης ε, παραμένει ότι ε, το περιθώριο έκθεσης ε, μπορεί να σημαίνει μεγάλο κίνδυνο κυρίως για καταναλωτές με μεγάλη έκθεση σε όλες τις ηλικιακέ ομάδες. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα τις ερωτήσεις σας. Uh, ευχαριστώ. Ο κύριος Φερστρέτερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά τα συμπεράσματα της ΕΦΣΑ, όπου η παρουσία του, των εστέρων MCPD και των εστέρων ε, γλυκιδόλης σε ραφιναρισμένα ε, φυτικά έλια δημιουργούσαν πρόβλημα υγείας. Γι' αυτό ακριβώς ξεκίνησε αμέσως η Κομισιόν συζητήσεις με τα κράτη-μέλη, ούτω ώστε να ληφθούν αυστηρά κανονιστικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία. Ε, Επίση, έγινε μια συζήτηση για να έχουμε αυστηρά τα όρια για τους εστέρες ε, γλυκιδόλης και τους εστέρες MCPD στα φυτικά έλαια. Καθώς και τα φυτικά έλαια που μπαίνουν στην αγορά για τους καταναλωτές, καθώς και τα φυτικά έλαια τα οποία χρησιμοποιούνται από, την ε, εταιρεία, από τις τροφίμων για να φτιάξουν τρόφιμα. Επιπλέον, όπως ακούσατε, υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία που συνδέεται με τη χρήση των εστέρων MCPD και των εστέρων γλυκιδόλης σε παιδικά γάλατα και γάλατα που τα παίρνουν σε μεγαλύτερες ηλικίε. Ε, για να προστατεύσουμε αυτή την ευάλωτη ομάδα πληθυσμού, η Κομισιόν σκοπεύει να θέσει αυστηρά όρια για τους εστέρες λυκηδόλη και τους εστέρες MCPD στα παιδικά γάλατα πρώτης ηλικίας και αυτά που παίρνουν τα παιδιά αργότερα, τόσο ώστε να υπάρχει υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας, καθώς και η ε, έκθεση των ε, νεογνών ε, που τρέφονται αποκλειστικά με παιδικό γάλα δεν δημιουργεί ουσιαστικό πρόβλημα υγείας. Επίσης η Τζέκφα σε σχέση με τους εστέρες 3 SCPD, MCPD έχει καταλήξει διαφορετικά συμπεράσματα από την ΕΦΣΑ και ακριβώς γι' αυτό η ΕΦΣΑ αποφάσισε να ξαναδεί την γνωμοδότησή της σε ό,τι αφορά τους εστέρες 3 ε, MCPD και να φτάσει σε τελικό συμπέρασμα μέχρι το τέλος του 2017. Γι' αυτό ακριβώς η Κομισιόν αποφάσισε να προχωρήσει με τα μέτρα σε ό,τι αφορά τους εστέλες γλυκιδόλες που είναι ε, γενοτοξικοί και καρκινογόνες, καρκινογόνοι με ανώτατα αυστηρά όρια για αυτούς τους εστές, καθώς και για τα ραφιναρισμένα φυτικά έλαια που μπαίνουν στην αγορά απευθείας για τον τελικό καταναλωτή, αλλά και τα φυτικά έλαια, τα ραφιναρισμένα που χρησιμοποιούνται από τους κατασκευαστές τροφίμων και από, ε, για αυτά που χρησιμοποιούνται στο παιδικό γάλα και στο παιδικό γάλα για μεγαλύτερες ηλικίες. Για τους εστέρες 3MCPD περιμένουμε τα αποτελέσματα αυτής της νέας ε, ε, επαναξιολόγηση της γνωμοδότησης και μετά από αυτό το αποτέλεσμα η Κομισιόν, ε, καμία καθυστέρηση, θα προτείνει μέγιστα όρια για τα φυτικά έλαια, ραφιναρισμένα φυτικά έλαια, παιδικό γάλα νεογνών και μεγαλύτερων παιδιών, ούτω ώστε να υπάρχει ψηλό επίπεδο δημόσιας υγείας. Ευχαριστώ. Thank you very much. Now I open the floor to the... Και τώρα δίνω το λόγο στους ευρωβουλευτέ. Σηκώστε το καρτελάκι σα, αν θέλετε να μιλήσετε παρακαλώ για το θέμα αυτό. Ο κύριος Λίζε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την εκπρόσωπο της ΕΦΣΑ αλλά και τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Προς την ΕΦΣΑ δεν έχω ερωτήσεις. Αυτό που μας είπε ήταν απόλυτα σαφή και η ΕΦΣΑ πολλές φορές επικρίνεται για το ότι κάποιοι κίνδυνοι δεν εκφράζονται με απόλυτη σαφήνεια. Εγώ δεν συμφωνώ, δεν συμμερίζομαι αυτή την κριτική. Πάντως και η ΕΦΣΑ το είπε με απόλυτη σαφήνεια ότι κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει έτσι ώστε να περιοριστούν αυτές οι ουσίες στη διατροφή για να μπορούμε πραγματικά να προσφέρουμε ασφάλεια στον καταναλωτή. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ την Κομισιόν. Κάνατε μία πρόταση για τη γλυκιδόλη. Τώρα, τι θα γίνει στη συνέχεια. Ε, υπάρχει μια επιτροπή που ασχολείται με το θέμα, ε, τι προτίθεται να κάνει η επιτροπή, ποιες είναι οι προθεσμίες και τι μπορούμε να κάνουμε εμεί ως κοινοβούλιο, έτσι ώστε οι πρώτες κομισιόν που κατά δική μου άποψη είναι τεκμηριωμένοι, πώς μπορούμε να στηρίξουμε την πρόταση αυτή. Ε, υπάρχει άραγε αντίδραση από κράτη-μέλη. Υπάρχουν ε, τεχνικά προβλήματα που να προβάλλονται κατά της πρότασης. Και πώς τα αξιολογείτε όλα αυτά. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω τι ακριβώς θα συμβεί συγκεκριμένα, πότε, πώς και πώς αξιολογείτε τις ε, πλειοψηφικές σχέσεις έτσι ώστε στο Κοινοβούλιο να μπορούμε και εμείς να εξάγουμε τα συμπεράσματά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. επειδή έγιναν προηγούμενες παρεμβάσεις, ε, ελπίζω να μην, δώσω, να μην πω κι εγώ τα ίδια. Άκουσα την Κομισιόν που είπε για αυτή την ανησυχία, την οποία συμμερίζομαι σε ό,τι αφορά την ε, παρουσία επιμολυντών στα, ε, για την παραγωγή παιδικού γάλακτος. η, εθνική, γερμανική εθνική, ο γερμανικός εθνικός φορέας για την υγεία και το περιβάλλον έδειξε ότι στα δείγματα παιδικού γάλακτος έχουμε μεγάλες περιεκτικότητες σε 3 MCPD. Παρότι υπάρχει διαφοροποίηση από προϊόν σε προϊόν, γενικά υπάρχει υψηλή περιεκτικότητα. Η Κομισιόν θα κάνει κάτι. Μπορείτε να μας δώσετε μια ιδέα για το τι θα γίνει στη συνέχεια, ε, τι θα γίνει με τα δεδομένα, με το χρονοδιάγραμμα κτλ. Ούτως να δω τι θα κάνουμε για το θέμα αυτό. Άλλα δύο θέματα, πολύ σύντομα. Ε, επίσης, η γλυκιδόλη θεωρείται τοξική και καρκινογόνα τι πιστεύει η Κομισιόν και η ΕΦΣΑ για αυτό το θέμα και αν υπάρχουν μέτρα ή εθελοντικά μέτρα για να περιορίσουμε περαιτέρω την γλυκιδόλη ε, σε τρόφιμα, ε, στο φινικέλαιο και στα λίπη. Επίση, για την συνειδητοποίηση των καταναλωτών για αυτά τα θέματα. Πιστεύω ότι δεν τα ξέρουν αυτά οι καταναλωτοί. Ε, δεν ξέρουν την σημασία αυτών των επιμολυντών. Πώ του αποφύγει, ποια, ποιοι επιμολυντέ υπάρχουν κτλ. Η Κομισιόν σκοπεύει να προωθήσει κάποια πρωτοβουλία τόσο ώστε να αυξήσει τη γνώση των καταναλωτών για τα θέματα αυτά που αφορούν τους συγκεκριμένους επιμολυντέ για τους οποίους μιλάμε σήμερα. Ευχαριστώ. κυρία Γιούσο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την ΕΦΣΑ και την Κομισιόν για την παρέμβασή της για το θέμα του φινικελαίου που τουλάχιστον στη χώρα μου δημιουργεί κοινωνική ανησυχία. Χτυπάνε καμπανάκια. Η Κομισιόν πότε θα πάρει μέτρα για να θέσει ανώτατα όρια. Και επίσης, σας έψα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Το πιο ανησυχητικό θέμα είναι τα παιδικά γάλατα, τα γάλατα που χρησιμοποιούν τα νεογνά αντί να θυλάζουν. Εκεί υπάρχει μεγαλύτερη ανησυχία για την παρουσία αυτών των επιμολυντών. Εάν τα όρια τα οποία χρησιμοποιούνται σε αυτά τα γάλατα για την παρουσία του 3-MCPD και 2-MCPD που υπάρχει και στο ραφιναρισμένο ε, φινικέλαιο. Ε, αυτά τα όρια είναι ενισχυτικά. Ξέρουμε ότι η δόση είναι αυτή που μετράει. Παραδείγματο χάρη, η, η, η παρίνη μπορεί να είναι είτε θανατηφόρα ή μπορεί να σώσει τη ζωή κάποιου, ανάλογα με τη δόση που, στην οποία χρησιμοποιείται, η επαρίνη. Η δόση που χρησιμοποιείται είναι ανησυχητική, γιατί έτσι νομίζει ο κόσμος. Οι δόσεις ε, και η περιεκτικότητα στα παιδικά γάλατα είναι σωστές, γιατί ο κόσμος ανησυχεί. Επίσης, ε, οι ποσότητε αυτών των επιμολυντών στο ραφιναρισμένο φινικέλαιο. Ε, είναι σωστή ή είναι ανησυχητική η δόση. Ε, ο κ. Καπούτο. σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, η σημερινή συζήτηση γίνεται μετά από μεγάλη περίοδο που ήταν περίοδος εγκυμοσύνης μέχρι να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ λοιπόν την ΕΦΣΑ που επιβεβαίωσε σήμερα ε, τη μελέτη την οποία είχαμε αναθέσει πριν από ένα χρόνο και σε αυτή τη μελέτη γίνεται αξιολόγηση τριών τοξικών ουσιών που διαμορφώνται κατά τη διάρκεια βρίσματος ε, σε πολύ ψηλές ε, θερμοκρασίες. Μιλάμε για τη γλυκιδιόλη και για τις ουσίες Το 2 και το 3 MCPD, αυτές τις τρεις ουσίες. Οι ποσότητες ε, όταν είναι πάνω από 6, 0,6 ε, ε, σε σχέση με τα φυτικά έλα, αυτό είναι ένα επικίνδυνο όριο. Βεβαίως το πρόβλημα δεν είναι στο φινικέλαιο, αλλά στον τρόπο με τον οποίο παράγεται σε υψηλές θερμοκρασίες για να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Το φινικέλαιο λοιπόν αντικαθιστά τα λύπη που υπήρχαν κατά το παρελθόν, γιατί είναι πιο ε, φθηνό, πιο οικονομικό. Όμως αυτό που κυκλοφορεί, το φινικέλαιο, δεν είναι ένα προϊόν που παράγεται σε χαμηλή θερμοκρασία και υπάρχει στις μερέντες, ε, στα κριτσίνια, σε ε, πάρα πολλά ε, τρόφιμα που δίδονται στα παιδιά και γι' αυτό λοιπόν δημιουργεί πρόβλημα κυρίως στην υγεία των παιδιών. Εγώ έχω κάνει μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέω ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν για να διαφυλαχθεί η υγεία των πολιτών. Μήπως θα πρέπει εντωμεταξύ να ξεκινήσει μια εκστρατεία ενημέρωσης. Θεωρώ ότι είναι σκόπιμο να ακούσουμε την ε, ε, άποψη που μου έστειλε η Επιτροπή που λέει ότι προτίθεται να παρουσιάσει στη μόνιμη Επιτροπή για τα φυτά ε, και για τις ζωοτροφές μέχρι το τέλος αυτού του έτους μέτρα κανονισμού τα οποία έχουν ως στόχο να παρουσιάσουν τους στέρες ε, γλυκυντόλης και τη μειουσία του MCPD στο λάδι και στα φυτικά έλαια και αυτά θα τα πράξει με στόχο να προστατεύσει καλύτερα την ανθρώπινη αξία, κυρίως ε, των μωρών που θυλάζουν και των πολύ μικρών παιδιών. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει προστασία των ανθρώπων, κυρίως όπως σας είπα των θυλαζών των μωρών και των πολύ μικρών παιδιών. Η Κομισιόν όμως δεν θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει ειδική εκστρατεία ενημέρωση όσον αφορά στη χρήση του φοινικέλαιου στα τρόφιμα. Από τον Αύγουστο του 2016 μέχρι σήμερα τίποτα δεν έγινε. Δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο. για αυτά που είχαν ελεγχθεί. Και εγώ πιστεύω ότι δεν χρειάζεται πια, δεν εξυπηρετεί το να αφήσουμε να περάσει και άλλος χρόνος, να γίνουν και άλλες μελέτες, ε, γιατί κατ' ουσίαν η κατάσταση είναι ξεκάθαρη. Θεωρώ ότι είναι παράλογο και μετά από την ε, μελέτη της ΕΦΣΑ, την οποία και θα ήθελα να ευχαριστήσω με αυτή την ευκαιρία να την ευχαριστήσω ε, γιατί επιβεβαίωσε όλα αυτά που πιστεύαμε. Μέχρι τώρα, με πάση περιπτώσει, δεν έχουν ληφθεί μέτρα από την Επιτροπή. Και αυτό που με θλίβει περισσότερο είναι ότι παρά την προφορική ερώτηση την οποία υποβάλαμε αρκετή εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι πολιτικές ομάδες παρόλα αυτά δεν θέλησαν να ε, οργανώσουν μία συζήτηση στην Ολομέλεια. Ελπίζω λοιπόν μετά από τη σημερινή συζήτηση να κριθεί ότι πλέον έχει νόημα να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, αν θέλετε, η συζήτηση στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δίνετε να συζητήσουμε με την ΕΦΣΑ και με την Κομισιόν για το θέμα αυτό. Είναι περίπτωνα να επαναλάβουμε αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Συνειδητοποιούμε ότι για τα παιδικά γάλατα, όταν μιλάμε για τα παιδικά γάλατα, το θέμα είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, καταλαβαίνετε. Και οι προθεσμίες θα πρέπει να είναι οι πιο αυστηρές δυνατές. Η ΕΦΣΑ μας έδωσε ένα χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της μελέτης που θα πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος του 2017. Εγώ κάνω έκκληση να μειωθεί αυτή η προθεσμία ή δυνατόν και η Κομισιόν να μπορέσει να παρέμβει το συντομότερο δυνατόν, ούτω ώστε να ρυθμίσει τα θέματα αυτά με τρόπο πολύ αυστηρό, να ρυθμίσει το θέμα των ανώτατων ορίων ε, του επιμολυντη 3 MCPD για να προστατεύσει τους Ευρωπαίους καταναλωτές. με πολύ θετική εγώ απέναντι σε αυτή τη μελέτη που είναι, μας δίνει μια σφαιρική εικόνα για την παραγωγή όλων των ελαίων, όχι ανακατηγορία. Γιατί, όπως υπόθηκε ξεκάθαρα, αυτό που είναι σημαντικό είναι η μέθοδος ραφιναρίσματος που χρησιμοποιείται όχι τόσο πολύ η πρώτη ύλη αυτή αυτή. Και είναι σαφές ότι θα πρέπει να μειώσουμε την παρουσία αυτών των επιμόλυτων που οφείλονται στην υψηλή θερμοκρασία. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο πολίτης για τα προβλήματα αυτά και είναι σημαντικό να γίνεται έλεγχος για τη μεθοδολογία ραφιναρίσματος, για τη μέθοδο ραφιναρίσματος. Το πρόβλημα δεν είναι η, μέθο... Ε, το πρόβλημα δεν είναι η πρώτη ύλη. Το θέμα είναι πώς ε, ραφιναρίζεται αυτή η πρώτη ύλη και πώς χρησιμοποιείται. Νομίζω ότι η προσέγγιση είναι σωστή, ισορροπημένη. Θα ήθελα όμως η προθεσμία να είναι λιγάκι πιο αυστηρή. Να παρεύουμε το συντομότερο δυνατόν. Για να μην συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε ε, αυτά τα, αυτούς τους επιμολυντές στα τρόφιμα που οφείλονται στις υψηλές θερμοκρασίες για να μπορέσει ο καταναλωτής να χειριστεί την ε, κατάσταση, να διαχειριστεί το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Η ξανά το λόγο και εν συνεχεία η Κομισιόν για να απαντήσει. Γεύσα πρώτη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, κοιτάξτε, όσον αφορά την ερώτηση της κυρίας Αγιούσα, θέλω να πω, είναι αλήθεια ότι η έκθεση των μωρών σε στέρες γλυκιδόλης ε, ε, μέσα από το παιδικό γάλα είναι πολύ μεγαλύτερη εκθεσή, κατά 10 περίπου φορές από ότι κρίνεται ανώδυνο και ακίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Άρα δηλαδή το να υπάρχουν αυτές οι ενώσεις στο παιδικό γάλα αυτό γίνεται για διατροφικούς λόγους, γιατί αυτό το γάλα μοιάζει πάρα πολύ στο γάλα του θυλασμού. Βέβαια αυτό ανησυχεί, ανησυχεί για την ε, ε, διατροφή των μωρών που χρησιμοποιούν αυτό το παιδικό γάλα, αυτή τη μορφή παιδικού γάλακτος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούστηκε μία ερώτηση προς την Κομισιόν για το χρονοδιάγραμμα. Υπάρχει διαφορετικό χρονοδιάγραμμα ε, για τους αστέρες γλυκιδόλης που κατά την άποψη της ΕΦΣΑ ε, δεν θα πρέπει να ξανανοίξει ως θέμα. Αντίθετα, πρέπει να ξανανοίξει το θέμα της, ε, του 3MCPD. Για τους εστέρες γλυκιδόλης έχουμε ολοκληρώσει τις τεχνικές συζητήσεις με τα κράτη-μέλη και σκοπεύουμε να υποβάλουμε μία κανονιστική πρόταση για μέγιστα όρια φυτικών ορίων ε, που τίθεται απευθεία στην αγορά για τον τελικό καταναλωτή, καθώς και τα φυτικά έλαια που χρησιμοποιούνται στατικό από τους κατασκευαστές τροφίμων, καθώς και αυστηρά ανώτατα όρια για το παιδικό γάλα νεογνών και μεγαλύτερων παιδιών. Σε μία από τις επόμενες μόνιμες επιτροπές θα τα προτείνουμε αυτά ή μετά την εσωτερική διαδικασία διαβούλευσης της Κομισιόν θα, το, θα κάνουμε αυτές τις προτάσεις. Το σχέδιο είναι να υποβληθεί στην ε, μόνιμη επιτροπή λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές ή αμέσως μετά. Είναι ένα μέτρο το οποίο εντάσσεται στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, που σημαίνει ότι μετά την γνωμοδότηση τη μόνιμη επιτροπή στα πλαίσια τη Επιτροπολογία, το μέτρο θα υποβληθεί στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για έλεγχο ε, επί τρει μήνε και σε εκείνη τη φάση θα υπάρχει και η δυνατότητα να ακουστούν και οι απόψει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί αυτών που προτείνει η Κομισιόν για να εξασφαλίσει την προστασία της δημόσιας υγείας. Σε ό,τι αφορά το θέμα που θέσατε για το πώς θα εκπαιδεύσουμε τον καταναλωτή για αυτό το πρόβλημα, η παρουσία αυτών των εστέρων της μονοχλωροπροπανοδιόλης και των εστέρων γλυκοδιόλης στα φυτικά έλαια γίνεται κατά τη διάρκεια ε, ραφιναρίσματος των φυτικών ελαίων. Αντίθετα με άλλους επιμολυντές ε, κατά τη διάρκεια της κατεργασίας, ε, το, μαγείρεμα δεν επηρεάζει και δεν εμφανίζει αυτούς τους εστέρες, είτε γλυκοδιόλης ή μόνο χλωροπροπανοδιόλης. Μόνο ραφινάρισμα εμφανίζονται. Αυτό το ε, θέμα έχει εντοπιστεί. Έχουν ληφθεί κάποια θελοντικά μέτρα από τον κλάδο ραφιναρίσματος για να μειωθεί η παρουσία των εστέρων γλυκοδιόλης και των εστέρων 3-MCPD ε, στα ραφιναρισμένα φυτικά έλαια. Κατά τη γνωμοδότηση, στη γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ υπάρχει σοβαρή μείωση για τους, εσ... για τους εστές Όμως είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε αυστηρά κανονιστικά μέτρα ε, για να εξασφαλίσουμε την προστασία της υγείας. Ε, το λέει Επίσης συμφωνούμε με την ανησυχία που προκαλεί παρουσία αυτών των ουσιών στο παιδικό γάλα νεογνών και μεγαλύτερων παιδιών και γι' αυτό στην κανονιστική πρόταση που θα υποβάλουμε προς ψηφοφορία στην μόνιμη επιτροπή σε κάποια από τις επόμενες φάσεις επιτροπολογίας ε, θα προτείνουμε αυστηρά ανώτατα ε, όρια για τα παιδικά γάλα νεογνών και μεγαλύτερων παιδιών. Τώρα, σε σχέση με αυτά που ρώτησε ο κ. Καπούτο, η Κομισιόν είχε την πρόθεση να, βάλει, να υποβάλει αυτή την κανονιστική πρόταση ε, μέχρι τα τέλη του 2016 με βάση την πρόταση της ε, Επιτροπής του Μαΐου του 2016. Αλλά ενώ είχαμε προχωρήσει τις συζητήσεις, συνειδητοποίησαμε ότι η Τζέκφα, ε, η, επιτροπή, η Κοινή Επιτροπή του ΠΟΕ, θα κάνει και αυτή μια έρευνα για να υπάρξει μια διεθνή διάσταση και γι' αυτό περιμέναμε την αξιολόγηση της Τζέκφα e για να δούμε αν θα ευθυγραμμίζεται με την αξιολόγηση της ΕΦΣΑ ούτως ώστε να προχωρήσουμε με την κανονιστική πρόταση. Ε, σε ό,τι αφορά τους αστέλες γλυκιδόλης, όπως ακούσατε, δεν υπάρχουν μεγάλες ε, αποκλήσεις απόψεων της Τζέκφα e και της ΕΦΣΑ, γι' αυτό ακριβώς ε, συνεχίσαμε αμέσως τις συζητήσεις με τα κράτη-μέλη. Και όπως είπα, Ολοκληρώσαμε και σε τεχνικό επίπεδο τη διαδικασία και τώρα θα υποβάλουμε την πρόταση τους επόμενους μήνες για τελική οθέτηση από την Κομισιόν. Σε ό,τι αφορά τους αστέρες 3 ε, MCPD, η Κομισιόν πιστεύει ότι το συντομότερο δυνατόν θα πρέπει να μάθουμε το αποτέλεσμα μετά την αναθεώρηση από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας των Τροφίμων και όταν ε, καταλήξει συμπέρασμα η ΕΦΣΑ, αμελητή θα προτείνουμε κανονιστικά μέτρα για τους εστέρες 3 MCPD στους, στα φυτικά έλαια, στο παιδικό γάλα νεογνών και λίγο μεγαλύτερο παιδιών, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας. Ειδικά προστασίας της υγείας των ε, πολύ μικρών παιδιών και παιδιών. Όπως είπε η κυρία Γκαρντίνη, το βασικό πρόβλημα είναι το πρόβλημα της μεθοδολογίας. Η μεθοδολογία μπορεί να μας βοηθήσει για να μειώσουμε την παρουσία αυτών των επιμολυντών ε, και η βιομηχανία μεταποίησης και ραφιναρίσματος θα πρέπει να εφαρμόσει μεθοδολογίες ούτω ώστε ε, οι εστέρες ε, γλυκιδόλης και οι εστέρες 3-MCPD να είναι όσο να τον λιγότεροι σε τα φυτικά έλαια και στο παιδικό γάλα. Ο κύριος Καπούτο. Σύντομα παρακαλώ όμως. Κοιτάξτε, θα ήθελα να ευχαριστήσω για τις απαντήσεις που μας δώσατε. Θα ήθελα μόνο να κάνω μια διευκρίνηση. Κοιτάξτε, και εμένα μου κοστίζει σε σχέση με αυτούς, αυτή την πρόοδο που υπάρχει ε, στο ραφινάρισμα του φινικέλαιου. Όμως πρέπει να σας πω ότι δεν συμφωνώ με αυτό που είπατε σχετικά με τα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούμε καθημερινά στη μαγειρική μας. Ε, διότι το πρόβλημα υποτίθεται ξεκινάει από, την, ε, ε, από το ραφινάρισμα, αλλά όταν μια νοικοκυρά αγοράζει προϊόντα είναι ήδη ραφιναρισμένα. Το θέμα, αν το θέμα είναι να έχουμε συνειδητούς καταναλωτές. Εγώ πιστεύω ότι και από επιστημονική άποψη θα πρέπει να προσπαθούμε να ενημερώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τους καταναλωτές. Πολύ ωραία λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Έκλεισε η συζήτηση. Ήταν και το τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Θα τα ξαναπούμε. Στις 29 Μαΐου ε, προβλέπεται να είναι η επόμενη συνεδρίασή μας. Ευχαριστώ πολύ.